Possiamo dare inizio? Dobbiamo andare molto rapidi. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Αλλάζουμε τη σειρά των ψηφοφοριών για να επιτρέψουμε στην έκθεση Γκαρόνα να ψηφίσουν οι συνάδελφοι που πρέπει σε άλλη επιτροπή. Δεν έχουμε ακόμα τον τελικό κατάλογο ψηφοφοριών για την έκθεση Καρών. Πάμε στο σημείο 10 τροποποίηση του κανονισμού 1698 του Συμβουλίου όσον αφορά κάποιες ε, διατάξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση για κάποια κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες ή που απειλούνται με μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά την οικονομική τους ε, σταθερότητα, χρηματοοικονομική τους σταθερότητα. Ε, θέλουμε να προχωρήσει γρήγορη έκθεση για να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα κάποιων κρατών μελών. Ήδη ανακοινώθηκε πριν από λίγο συμφωνία με το Συμβούλιο πάνω σε αυτό. Αυτό που ψηφίζουμε σήμερα σχετικά αφορά την έκθεση αυτή για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα είναι η τελική νομοθετικού περιεχομένου έκθεση. Άρα πάμε στην Ολομέλεια κατευθείαν με την επιτευθύσα συμφωνία με το Συμβούλιο. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει αλλαγή να προσθέσουμε κάτι. Συζητήσαμε επανειλημμένο το θέμα με τον Διευθυντή της Γενικής Διευθύνσεως Άγκρη, Λορέτα Μαρίνο, που διευκρίνησε και ξεκαθάρισε όλα τα σημεία τα επίμαχα τα οποία θίγησαν και διασκεδάστηκαν ανησυχίε κάποιων κρατών μελών. Άρα θα έλεγα ότι δεν, έχουμε, δεν χρειάζεται να χρονοτριβήσουμε άλλο και μπορούμε να προχωρήσουμε στον κατάλογο ψηφοφοριών. Κατάλογος ψηφοφοριών. Δεν χρειάζεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μπορούμε να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που απέσυραν τις τροπολογίες για να μας επιτραπεί έτσι μία έγκριση ε, ταυτόχρονα με το Συμβούλιο του ώστε να υιοθετηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται το νέο νομοθετικό κείμενο. Συμφωνείτε, μπορούμε να ψηφίσουμε συνολικά. Δεν χρειάζεται η κάρτα τώρα, Λουίς, να ψηφίσουμε στο σύνολο, έτσι. Γενικά, ψηφίζουμε λοιπόν στο σύνολο συνολικά τις τροπολογίες που συμφωνήθηκαν με το Συμβούλιο. Ποιος υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνονται. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους και τώρα πάμε κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το νομοθετικό κείμενο, αλλά επίσημα θα πρέπει να ψηφίσουμε την νομοθετική πρόταση που τροποποιήθηκε επίσης υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται αυτά για την τυπική διαδικασία. Ευχαριστώ όλους. Μπορούμε τώρα στα γρήγορα να πάμε στην έκθεση Καρόνα για να επιτρέψουμε στους συναδέλφους Λαδία και σε άλλους να πάνε να ψηφίσουν στην άλλη επιτροπή που πρέπει να πάνε. Εντάξει, λοιπόν, σημείο 12 της ημερήσιας ε, διάταξης για να αποφύγουμε Πώ θα αποφευθεί η σπατάλη τροφίμων στατικέ για τη βελτίωση αποτελεσματικότητα τη τροφική αλυσίδα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισηγητή ο κ. Σαλβατόρε Καρόνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίζουμε μια έκθεση σημαντικότατη αυτή για τη σπατάλη τροφίμων και τι στατικέ για τη βελτίωση τη αποτελεσματικότητα τη τροφική αλυσίδα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποβλήθηκαν 88 τροπολογίες που επεξεργάστηκε ο εισηγητής και κατέληξε σε έξι βαστικές τροπολογίες ε, για να ψηφίσουμε. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ, η κυρία Κοράτσα Μπίλντ είναι εδώ μαζί μας και την ευχαριστώ γι' αυτό. Μας έδωσε μια γνωμοδότηση, τέσσερις παράγραφοι θα ψηφιστούν, ενώ το υπόλοιπο κείμενο, δώδεκα παράγραφοι, θα σου δώσω το λόγο, τώρα τελειώνω, κυρία Άγνιο, δεν χρειάζεται να συνεχίσει να χτυπά τα χέρια. Θα σα δώσω το λόγο όταν τελειώσω. Λοιπόν, 12 παράγραφοι καλύπτονται από την εισήγηση. Λοιπόν, η Επιτροπή ΕΜΒΗ ψήφισε τη γνωμοδότησή τη μόλι εχθέ. Οπότε ο κατάλογο ψηφοριών διενεμήθη και μπορούμε στο τέλο να ψηφίσουμε. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καρόνα, ο κύριο Σανιού ζήτησε το λόγο. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, έχω ένα τεχνικό πρόβλημα. Η φωνή σα Πρόεδρε, έρχεται, ακούγεται πάρα πολύ δυνατά και δεν ακούω τη φωνή των διερμηνέων. Διαρωτώ με και οι άλλοι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Θα... Οι τεχνικοί θα κάνουν τις δέσεις προσαρμογές. θα ξεκινήσουμε το μεταξύ. Ο κύριος Καρόνα έχει το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και όλος ιδιαίτερος τον συνάδελφο Λαβία, διότι πιστεύω ότι πάρα πολύ γρήγορα κατάφερε αυτή η Επιτροπή ε, να καταλήξει σε μια έκθεση σημαντικότατη που έχει συνέπειε όσον αφορά και την κοινή ε, γνώμη ε, που δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα διότι το θέμα είχε υποτιμηθεί επί μακρόν Και με την ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια πιστεύω ότι ανοίγει μια εποχή πάρα πολύ σημαντική και σημαντική και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Ευχαριστώ κύριε Καρόνα και τώρα θα πρέπει να έχετε εδώ τον κατάλογο των ψηφοφοριών, πρέπει να έχετε όλη αυτή, να έχετε όλη αυτό το κατάλογο. Ξεκινάμε λοιπόν τις ψηφοφορίες μας. Λοιπόν, Ξεκινάμε τη ψηφοφορία όσον αφορά την τροπολογία 1. Ανοιχτή ψηφοφορία λοιπόν. Ελεκτρονική ψηφοφορία μάλλον λέει ο Πρόεδρος. Non ho C'è un, voto in più per il e. Ok? Bene. Dichiaro la votazione. ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν. Προχωρούμε. Τροπολογία 2. Στο 2 ξεκινάμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στο σημείο 3. Down Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται. Τροπολογία 3. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 4. Αιτιολογική σκέψη 4. Λέει ο πρόεδρος είναι τροπολογία 4. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Chiusa la votazione. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία για την 7. Πέρας. Τροπολογία 7. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία για την 8. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. 12 και 13 είναι ταυτόσιμες. Πάμε στη 14, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 14. 14. Ψηφίσατε όλοι για 14, πέρας για τη 14 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη 15, άρχεται η ψηφοφορία για την 15. Πέρας ψηφοφορία για 15 εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για 16. Ψηφοφορία για την ε, τροπολογία 16. Πέρας Ψηφίζουμε τη 17. Εγκρίθηκε η 16. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 17. Ψηφίσατε όλοι για τη 17. Πέρα ψηφοφορία εγκρίνεται. 18. Νεντατσέβα. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 18. Άρχεται. πέρας Για τη 18 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη 19. Άλουαντ Γκουλάρ, άρχεται η ψηφοφορία για τη 19. Πέρας ψηφοφορίας για τη 19, εγκρίνεται. 20. Άρχεται η ψηφοφορία για την 20. Πέρας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 21. Άρχεται η ψηφοφορία για την 21. 21. Πέρας ψηφοφορίας για την 21. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 22. Μαγκίνες, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας για την 22, η οποία εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην ΙΜΚΟ 5. Ψηφίζουμε λοιπόν τη γνωμοδότηση Επιτροπής ΙΜΚΟ 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται πέρας για την ΕΜΚΟ 5 που εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 23. Άρχεται η ψηφοφορία για την 23. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Άρχεται η ψηφοφορία για την 24. Η 24. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται. Πάμε στην 25. Ψηφίζουμε την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26. Άρχεται η ψηφοφορία για την 26. Πέρας της ψηφοφορίας για την 26. Εγκρίνεται. 27. Άρχεται η ψηφοφορία για την 27. Μαγκίνες. 27. Εγκρίνεται. Πέρας ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 28. Μπεκάλι. Άρχεται η ψηφοφορία για την 28. Η 28 πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και έχουμε την 29 κοράτσα Μπίλτ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 29. Τροπολογία 29 άρχεται η ψηφοφορία πέρας αυτής απορρίπτεται. Απορρίπτει 29. Πάμε στην 30. Νταντέν. Άρχεται η ψηφοφορία για την 30. 30. Πέρας. Για την 30. Η οποία απορρίπτεται. Και αυτή. Ψηφίζουμε την 31. Άρχεται η ψηφοφορία για την 31. Άρχεται η ψηφοφορία. 31. Πέρας Απορρίπτεται και 31. 32. Ψηφίζουμε την 32. Ταραμπέλα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία στην 32. Εγκρίνεται. 33. Νικουλέσκου. 33. Πέρας εγκρίνεται 33, 34, 34. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται και αυτή. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ΙΜΚΟ 3. Ψηφίζουμε την τροπολογία της Επιτροπής ΙΜΚΟ 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Μετά πάμε συμβαστική 1. Συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική 1. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας η οποία εγκρίνεται. Η συμβαστική 1 εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 39. Άρχεται η ψηφοφορία για την 39. Πέρας ψηφοφορίας. Πάμε στη 40 λέει ο Πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 40. Ρολάντας Πάξας. Πέρας ψηφοφορίας για τη 40. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 41. Ράρες Λούσαν Νικουλέσκου. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 42. Σε τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία το πρώτο τμήμα τη 42. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο τμήμα της 42. Δεύτερο τμήμα της 42 ψηφίζουμε. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει πλειοψηφία υπέρ. Το δεύτερο τμήμα της 42 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη 43. Κοράτσα Μπίλτ. Σωστά. Όχι. Όχι, όχι, όχι. όχι. Η 42 όχι. Πάμε στην τροπολογία 45. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 45. 45, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 46. 46. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 46. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε φορή τη 46, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη 47, μάνερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 47, μάνερ. Πέρας. Απορρίπτεται. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Τέλος πάω. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πού είμαστε? 48 είναι το επόμενο σημείο. Άρχεται η ψηφοφορία στην τροπολογία 48 είμαστε. πέρα τροπο, ε, ψηφοφορίας για τη 48 εγκρίνεται. 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 49. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 51 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία τροπολογία 51 Μαγκίνες. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 51. 52 άρχεται η ψηφοφορία για την 52. 52. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 53 Άρχεται η ψηφοφορία, τροπολογία 53. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική 2. Συμβιβαστική 2, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 61, κοράτσα Μπιλτ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 61. Bene, approvato. Καλώς εγκρίνεται. 62. Άρχεται η ψηφοφορία για την 62. 62, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 62. 63. Νικουλέσκου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας για την 63. Εγκρίνεται. 64. 64. Πέρας Απορρίπτεται 64. 65. Άρχεται η ψηφοφορία για την 65. Πέρας. Εγκρίνεται. 66. Ταραμπέλα. Άρχεται η ψηφοφορία. 66. Τροπολογία 66. Πέρας. Εγκρίνεται συμβιβαστική 3 που συμπεριλαμβάνει και την ΙΜΚΟ, συμβιβαστική 3. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία ΙΜΚΟ 15. Άρχεται η ψηφοφορία για την ΙΜΚΟ 15. Πέρας. Εγκρίνεται η ΙΜΚΟ 15. Συμβιβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβιβαστική 4. Πέρας. Εγκρίνεται. 76. Ταραμπέλα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 76. Πέρας. Εγκρίνεται, ψηφίζουμε τη συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική 5. Εγκρίνεται. Μάλιστα. Εγκρίνεται η συμβαστική 5. Πάμε στην ΙΜΚΟ 12 τώρα. ΙΜΚΟ 12 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 6. Πέρας. Συμβιβαστική 6 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 88 Πάξας. Άρχεται η ψηφοφορία για την 88. Εγκρίνεται και αυτή. Και τώρα ψηφίζουμε Προσοχή τον κατάλογο ψηφοφοριών που αλλάζει. ΙΜΚΟ 1. Άρχεται η ψηφοφορία επί της ΙΜΚΟ 1. Πέρας. Εγκρίνεται. Προσοχή τώρα. ΙΜΚΟ 4 πάμε. ΙΜΚΟ 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας για την ΙΜΚΟ 4. Uh, ε, Να διευκρινίσω τι ψηφίζουμε με τις τελευταίες ψηφοφορίες. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ δεν απεδέχθη τη δική μας σειρά ψηφοφοριών που βλέπετε στον κατάλογο ψηφοφοριών. Γι' αυτό προσέξτε τα νούμερα, τους αριθμούς. Διότι είναι μόνο εκείνα που πέρασαν από την ΙΜΚΟ σήμερα το πρωί. Διαβάζω με πολύ προσοχή τον αριθμό. Μην κοιτάτε τη σειρά του καταλόγου που έχετε στον πίνακα σήμερα το πρωί άλλαξε. Καλώς ψηφίσαμε την ΙΜΚΟ 1 και την ΙΜΚΟ 4. Τώρα λοιπόν τελείωσε αυτή η ψηφοφορία έτσι. Α, ξεκινάμε την ψηφοφορία επί της ΙΜΚΟ 8. 8 ΙΜΚΟ. Άρχεται η ψηφοφορία. ΙΜΚΟ 8. Προσοχή στους αριθμούς. Πέρας ψηφοφορίας. ΙΜΚΟ 8 λοιπόν εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην ΙΜΚΟ 10. ΙΜΚΟ 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας. Η 10 εγκρίνεται. Πάμε στην ΙΜΚΟ 13. 13. ΙΜΚΟ 13. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας ΙΜΚΟ 13 που εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την ΙΜΚΟ 17, 1-7, ΙΜΚΟ 17. Άρχεται η ψηφοφορία για την ΙΜΚΟ 17. Ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας για την ΙΜΚΟ 17. Εγκρίνεται και αυτή. Τελευταία τροπολογία της Επιτροπής ΙΜΚΟ είναι η ΙΜΚΟ 18. ΙΜΚΟ 18, 1-8, 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται και αυτή. Πολύ καλά. Πάμε στροπολογίε στην, ε, τροπολογία Επιτροπή Επιτροπής Περιβάλλοντος. Επιτροπή Περιβάλλοντος, τροπολογίες Επιτροπής αυτής. Έτσι. Ξεκινάμε από την NV4. Άρχεται η ψηφοφορία για την NV4. Πέρας ψηφοφορίας. Η NV4 εγκρίνεται. NV5. Άρχεται η ψηφοφορία. NV5. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται η NV5. nv 20 Άρχεται η ψηφοφορία για την nv 20 NV20. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται η nv 20 Ψηφίζουμε τώρα την nv 32 Άρχεται η ψηφοφορία. MV32. Πέρας ψηφοφορίας για την MV32. Εγκρίνεται. Πάμε στην MV33. Άρχεται η ψηφοφορία. MV33. MV33. Ψηφίσατε όλοι την εν λόγω τροπολογία. Πέρας. Απορρίπτεται η MV33. MV50. Άρχεται η ψηφοφορία. MV50. Πέρας για την MV50 η οποία και εγκρίνεται. MV57 MV57 ψηφίσατε όλοι για την 57 περας εμβι MV57 εγκρινεται εμβι MV70. Άρχεται η ψηφοφορία για την εμβι 70 κοντά. Πέρας για την εμβι 70 η οποία εγκρίνεται. MV88 άρχεται η ψηφοφορία MV88 πέρας εγκρίνονται. Έμβη 91 και τελειώνουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος με αυτήν. Έμβη 91 άρχεται η ψηφοφορία. Έμβη 91 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματος που τροποποιήθηκε. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία όσον αφορά την πρόταση ψηφίσματος που τροποποιήθηκε. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα τελειώσαμε. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο Καρόνα. Μπορούν να πάνε να ψηφίσουν οι συνάδελφοι. Πάμε στο σημείο 11 που αφορά την προμήθεια των ερωτικών ε, προϊόντων. Ο Ιωσέ Μπουβέ έχει το λόγο. Η αλυσίδα προμήθεια των γεωργικών εισρώων, διάθεση και προεκτάσει. Εδώ έχουν παρουσιαστεί 229 τροπολογίε και έχουμε τρει συμβαστικέ τροπολογίε. Ο κύριο Μποβέ λοιπόν έχει το λόγο και ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι παρόντες. Ο Γιωζέ έχει το λόγο. Δεν θα κάνω δηλώσει στη συζήτηση αυτή. Δουλέψαμε σκληρά. Υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες διότι οι πάντες ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Κατορθώσαμε να καταθέσουμε τρεις συμβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό διότι υπάρχουν ποικίλε απόψεις Πρέπει να σεβαστούμε την ποικιλομορφία των τροπολογιών. Σας καλώ λοιπόν να ψηφίσετε υπέρ του γενικότερου συμφέροντος των αγροτών, διότι ακριβώς αυτούς προσπαθούμε να προστατεύσουμε, ούτως ώστε να ε, ε, ούτως ώστε να μην, το, το, κόστο, το υψηλό κόστος της παραγωγής να μην τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν την δραστηριότητά τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χωσέ. Ξεκινάμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Θα προσπαθήσω να προχωρήσω στο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν, ε, έχουμε πολλές ψηφοφορίες πρέπει να κάνουμε. Ξεκινάμε με την τροπολογία 89. Μαγκίνες. Άρχεται η ψηφορία για την 89. Πέρας για την 89. η οποία εγκρίνεται. 90. 90, τροπολογία 90, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Adesso andiamo al 92, Lion ed altri. Votazione 92, Lion και άλλοι. Άρχεται η ψηφοφορία για την 92. Ops. Chiuso. 90... Πέρας 92. Εγκρίνεται. 93. Άρχεται η ψηφοφορία με την 93. Lion και άλλοι. Άρχεται η ψηφοφορία 93. Πέρας. Εγκρίνεται η 93. 94. Άρχεται η ψηφοφορία για την 94. Πέρας. Η 94 εγκρίνεται. 95. Άρχεται η ψηφοφορία για την 95. 95. Πέρας. Εγκρίνεται η 95. 96. Ε, Νίκολσον. Άρχεται η ψηφοφορία. 96. Πέρας. Δανέλης. Σπύρο, να σε βλέπω. Ε, λοιπόν, εγκρίνεται 96. 97. Άρχεται η ψηφοφορία για την 97 πέρας για την 97. Η 97 απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 98 σε δύο ξεχωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της 98. Πέρας. Το πρώτο τμήμα της 98 μαγκίνης εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα ψηφίζουμε της 98. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα Δεύτερο τμήμα ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 99. Άρχεται η ψηφοφορία για την 99. Πέρας απορρίπτεται. Πάμε στην 100. Άρχεται η ψηφοφορία για την 100. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας Απορρίπτεται 100. 101. Άρχεται η ψηφοφορία. 101. 101. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 109 στην επόμενη σελίδα. 109. Ψηφίσαν όλοι. Πέρας εγκρίνεται 109. 110. Άρχεται η ψηφοφορία για την 110. 110. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 1. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 1. Ψηφίσατε όλοι εγκρίνεται. 117 Πατράου 117 Ψηφίσατε όλοι την 117 πέρας εγκρίνεται 118 Τελάνος. άρχεται η ψηφοφορία 118 Ψηφίσατε όλοι την 118. Πέρας. Εγκρίνεται. 119. 119. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 120. 120. Ψηφίσατε όλοι την 120. Εγκρίνεται. 121 Δανέλης. 121. Ψήφισαν όλοι. 121 εγκρίνεται. 122 Λάιον και άλλοι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι την 122. Πέρας. Εγκρίνεται η 122. 123. Όχι. Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. 126. 126. Άρχεται η ψηφοφορία για την 126. 1, 2, 6. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 127. Άρχεται η ψηφοφορία για την 127. Πέρας. 127. Εγκρίνεται μάλλον. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα. Ε... Πάμε. 130. 130. 130. Γέγκλε και Ντες. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 131. 131. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 132. Άρχεται η ψηφοφορία. 132. Πέρας. Απορρίπτεται. 133. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 133. Απορρίπτεται και αυτή. Poi andiamo al 134, Dantin, aperta la votazione sul 134. 134 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία για 134, πέρας εγκρίνεται. 135. Άρχεται η ψηφοφορία για την 135. Votazione chiusa, 135 approvato. Εγκρίνεται 135. 137. Ψηφίζουμε την 137. Πέρας. Εγκρίνεται. 138 Μακίνες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας για την 138 που εγκρίνεται. Πάμε στην 140. Άρχεται η ψηφοφορία. 140. Πέρας για την 140. Εγκρίνεται. 142, Λαβία, 142, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται 142. 143 Κόστιγκερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 143. 145. Άρχεται η ψηφοφορία για την 145. 145 Γκλατφέλντερ απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 146 Φοντάνα. Άρχεται η ψηφοφορία 146. Πέρας. Απορρίπτεται. 147. Άρχεται η ψηφοφορία για την 147. 147. Πέρας εγκρίνεται 148 Δες και άλλοι, άρχεται η ψηφοφορία για τα 148 ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται 149 down 10 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. Νταντέν δεν χάνει τίποτε. ούτε. 150 Νικουλέσκου, άρχεται η ψηφοφορία, 150. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, 150 απορρίπτεται. 151. Άρχεται η ψηφοφορία για την 151. Γέγκλε. Ψήφισαν όλοι. Ναι. Πέρας. Εγκρίνεται. 152. Άρχεται ψηφορία για την 152. Πέρας. Μεγάλη πλειοψηφία κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. 153. 153 ψηφίσατε όλοι. Γκλάτφέτερ απορρίπτεται. Adesso votiamo il 154. 154. η ψηφορία για την 154. Ψηφίσατε όλοι. Λάιον και άλλοι. 154. Απορρίφτεται 154. 155. Ντελάνζ. 155. Ψηφίσατε όλοι την 155. Πέρας Εγκρίνεται 155. Πάμε στην 157 Gladfelder. Άρχεται η ψηφορία την 157. 157. Πέρας για την 157. Απορρίπτεται μάλλον. Και Νταντένα 158 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται πέρας 158. Δαντέν εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται. Α, α, να και μια φορά. Νταντέν, εδώ έχασε. 159. Άρχισε ψηφοφορία. 159, λοιπόν, πέρας. 159 εγκρίνεται. 162 μορβάει. 162 μορβάει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας η 162 απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Συμβιβαστική 2 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αλλάζουμε σελίδα και πάμε στην 175. 175. Ντελάουνς και άλλοι. Άρχεται η ψηφοφορία. 175. Πέρας. Εγκρίνεται. 177. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 177.

Η 178 εγκρίθηκε. Τελειώσαμε με αυτήν και πάμε στην 179 γέγκλε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 179. 179 που νομίζω ότι εγκρίνεται και η 179. Για να δούμε. Ναι, πέρασε αυτή. Πάμε στην 180. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 180. 180. πέρασε. Εγκρίνεται λοιπόν και 180. 181. 181. Εράνς Γκαρσία και άλλοι. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 181. Πέρας. Εγκρίνεται 182 Νίκολσον. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 182. 182 πέρας. Νομίζω ότι απορρίπτεται. απορρίπτεται. 183. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 183. 1, 8, 3. Πέρας. 183. Εγκρίνεται. 188. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 188. 188 Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 189. Άρχεται η ψηφοφορία. 189 Δανέλης. Πέρας. Απορρίπτεται 189. 190 Ρέιμερς. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 190. Πέρας. 190 εγκρίνεται. 192 μπεκάλι άρχεται η ψηφοφορία πέρας Απορρίψατε 192 Συμβιβαστική 3 άρχεται η ψηφοφορία επί της συμβιβαστικής 3 Ψηφίσατε όλοι, εγκρίνατε. Αλλάζουμε σελίδα και πάμε στην 207. Νικουλέσκο. 207. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 207. Πέρας. Απορρίπτεται 207. Και τώρα πάμε στη 208. 208 Νταντά. Πέρας. ο Ντατέν ξεχωρίζει από την ομάδα. Α, απορρίπτεται. Η 208. 209, Πάουλσεν και άλλοι. 209 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μεγάλη πλειοψηφία για την Αντιπρόεδρο Πόλσεν. Πάμε στην 211 τώρα. 211. Ψηφίσατε όλοι. 211 απορρίπτεται. 212. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 212. Πέρας επί της 212. Απορρίπτεται. 212. Πάμε στη 214. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 214. Πέρας. Εγκρίνεται. 216. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 216. Πέρας. Απορρίπτεται. 217 Σμιτ. Σμιθ μάλλον. 217. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 219. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 219. Μαγκίνες, θες να πεις κάτι? Είπατε, μάλλον, τι, ψηφίσαμε προηγουμένως. Πού είμαστε, σε ποιο σημείο, τι ψηφίζουμε. 219. Καλώς, ευχαριστώ. Στο Γιάννοφ Μπίνεφ. Άρχεται η ψηφοφορία από τις 219 στο Γιάννοφ Μπίνεφ. Πέρας. Απορρίπτεται. 220 Λούλινγκ. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. 220 της κυρίας Λούλινγκ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται και αυτή. 221 Εράν Σκαρθία και άλλη Άρχεται η ψηφοφορία επί της 221. 221 που εγκρίνεται. 222 Ρούμπιξ. 222 εγκρίνεται. 223 άρχεται η ψηφοφορία. 223. Πέρας. Εγκρίνεται. 224 Ντελάνζ, άρχεται η ψηφοφορία. 224. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας για τη 224, η οποία εγκρίνεται 225 Άρχεται η ψηφοφορία επί της 225. Reimers εγκρίνεται. 226. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 226. Πέρας. Εγκρίνεται. 227 Ρούμπιξ. Πέρας επί της 227 εγκρίνεται. Λαβία 228 πέρας ψηφοφορία, 228 εγκρίνεται. 229 άρχεται η ψηφοφορία. Φοντάνα 229 πέρας εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις τώρα. Πάμε στην τροπολογία 8, Άλβες. Άλβες 8. Πέρας εγκρίνεται η τροπολογία 8. Τροπολογία 9, Κόστιγκερ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10, άρχεται η ψηφοφορία για τη 10. 10, ψηφίσατε όλοι. Τροπολογία 10, πέρας, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, 11. Ψηφίσατε όλοι την τροπολογία 11. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12, Λάιον και άλλοι. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 13, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η τροπολογία 13 εγκρίνεται. Τροπολογία 14, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τροπολογία 15. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. 16. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. 17. Πέρας. Τροπολογία 17 εγκρίνεται. Τροπολογία 18 άρχεται η ψηφοφορία. 18. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 άρχεται η ψηφοφορία. Γιατί 19. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Considerando 21. Τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 22. Τροπολογία 23, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται 23. Τροπολογία 24, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτεται 24. Τροπολογία 25, άρχεται η ψηφοφορία για την 25, Κόστιγκερ, πέρας, απορρίπτεται. Α, εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Έκανα λάθος, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε την τροπολογία 26. 27, συγγνώμη, διευθύνω διερμηνέας. 27 ψηφίσατε όλοι. Η 27 εγκρίνεται. 28, Νίκολσον, άρχεται η ψηφοφορία. 28. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 29. Ψηφίσατε όλοι. 29. Πέρας εγκρίνεται. 30. Χεράνς Καρσία και άλλοι. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 30. Πέρας. Για την 30 εγκρίνεται. 31 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 33 Νταντέν, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται λοιπόν για την τροπολογία 33, πέρας Η τροπολογία 33 απορρίπτεται. Πάμε στην 34. Άρχεται ψηφοφορία επί της 39, 34. Ε, Πέρας για την 34. Εγκρίνεται. 38. 38 Νίκολσον. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία 38. 39 άρχεται η ψηφοφορία επί της 39 απορρίπτεται η 39 ψηφίζουμε τη 40 Δανέλη άρχεται η ψηφοφορία για τη 40 πέρας και η 40 απορρίφθηκε 41 Άρχεται η ψηφοφορία επί τη 41. Τροπολογία 41. Ψηφίσατε όλοι. Εράν Καρσία και άλλοι. Η 41 εγκρίνεται. 42. Κόστιγκερ. 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 43. Εράνς Καρσία. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 43. Πέρας. Εγκρίνεται. 48. Δανέλη. 44. Νικουλέσκου. 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Για τη 44. Πέρας. 45 Νίκολσον, άρχεται η ψηφοφορία. 45, πέρας, εγκρίνεται, 50. Δανέλης, dichiaro aperta la votazione sul recital G. Άρχεται λοιπόν η ψηφορία επί της 50, Δανέλη. Που αφορά την αιτιολογική σκέψη J λατινικό. Ψηφίσατε όλοι. Την 50 Πέρας. Απορρίπτεται. 51. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 51. Ε, 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Oui, oui, non, non. Sì, sì, 52, scusi. 52 non... 51 non c'è. Chiedo scusa, allora votiamo, apriamo, apriamo il voto sul 52 recital K Nicholson, aperta la votazione. 52, γιατί 52, 52. Votazione sul 52 ed è... Η 52 εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. 53, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας για την 53. Ed è Approvato 55. Λοιπόν, εγκρίνεται 55 τώρα. πέρα. για την 55 εγκρίνεται 57 ντες και άλλοι άρχεται ψηφοφορία για την 57 άρχεται πέρας 57 Approvato. 59. Εγκρίνεται 59 άλβες. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται επί της 59. Chiusa la votazione sul 59. E Εγκρίνεται. Πάμε στην 60. Ε, Μορβάη. Τροπολογία 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται η 60. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 61. 61 Κόστιγκερ. Πέρας. Εγκρίνεται η 61. 62. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 62. Νταντέν. Κιούσα, Πέρας εγκρίνεται 63 Μορβάη 63 άρχεται η ψηφορία πέρας 63 λοιπόν απορρίπτεται ψηφίζουμε την 60 No. Niente. 65 allora. O il 73? Sì. sì. 65 Gladfelder. 65 άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας για την 65. Απορρίπτεται. Και τώρα να, δώσω το λόγο στην κυρία Μαγκίνες που ζήτησε το λόγο για κάποια τροπολογία προφορική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να υπάρχει συνέπεια στο κείμενο προτείνω να αντικαταστήσουμε την, ε, τον όρο crop rotation ε, με τη λέξη crop diversification, διαφοροποίηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που είναι αντίθετος με αυτή την αλλαγή που προτάθηκε. Δεν ε, υπάρχει αντίρρηση. Ο Ζωζέ Μποβέ έχει κάτι να πει. Η αμυψή βιοπικιλότητα. Ε, ε, ε, θέλουμε να μείνουμε με απόλυτα συνεπείς με το συμβαστικό κείμενο. Σήμερα έχουμε ένα συμβαστικό κείμενο. Άρα πρέπει να το τηρήσουμε αυτό. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, λοιπόν, ψηφίζουμε την πρόταση της κυρίας Μαγκίνες. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι. Non ho capito, scusa, allora sono io che non ho capito. Eh. Κάτι δεν κατάλαβα. Είσαι υπέρ ή κατά, Ζωζέ. Υπέρ ή κατά της προφορικής τροπολογίας. Contre. Είμαι κατά, κατά. Υπέρ, αν παραμείνουμε με το κείμενο ως έχει στη συμβαστική 2. Αν κρατήσουμε το κείμενο της συμβαστικής 2. αλλάζουμε κάτι ενώ έχουμε το σύνολο των αλλαγών συμβαστική 2. Άρα τι, τι να αλλάξουμε τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Η ε, κυρία Μαγκίνες τώρα. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι ε, το οποίο διαφοροποιείται από το συμβαστική λύση. Η κυρία Μαγκίνες πρέπει αν η ίδια δέχεται ότι παραμένουμε εντός των πλαισίων του συμβιβασμού, εντάξει. Η κυρία Μαγκίνης έχει το λόγο. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κύριο Μποβέ ότι παραμένω στο, κείμενο του το συμβαστικό. Το διαβεβαιώνω. Ωραία, ξεκαθαρίστηκε μας το πλαίσιο συμβαστικής 2, άρα δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από πλευρά ουδένος, Άρα ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία που είναι η κυρία Μαγκίνε. Λοιπόν, ε, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Abbiamo chiuso. Peras. Εγκρίνεται λοιπόν. Προχωράμε. Votiamo il 73 Reimers, aperta il voto sull'emendamento 70. Τροπολογία 73 Reimers, άρχεται η ψηφοφορία για την 73 πέρας για την 73 απορρίπτεται ψηφίζουμε την 74 άρχιε ψηφοφορία Chiusa la votazione su 74 direi Πέρας εγκρίνεται η 74 75 τώρα όχι Eh sì, 75 eh τώρα 75 άρχεται ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας για την 75 απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 76 δες και άλλη. Άρχεται ψηφοφορία για την 76. Πέρας. Εγκρίνεται. E poi votiamo il 70. 79 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 79. Ντελάος και λύπη. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 79. 80. 80. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 80. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε. 82, 82 μαγκίνε, άρχεται η ψηφοφορία. 82. Πέρας. Εγκρίνεται 82. 83 τώρα. Όχι, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρο 87. 87. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 87. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα Νίκολσον, τροπολογία 1. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2. Άρχεται ψηφοφορία. Γιατί 2 πέρας εγκρίνεται. 3. Άρχεται η ψηφοφορία. τρία Πέρας. Εγκρίνεται. τέσσερα Πέρας. Μάλλον άρχεται η τέσσερα τέσσερα Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η τέσσερα 5. Άρχεται η ψηφοφορία για την 5. 5. Εγκρίνεται. 6. Μορβάει. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το κείμενο του ψηφίσματος, Μποβέ, ως τροποποιήθη ed è definitivamente approvata. Bene. Εγκρίνεται λοιπόν το κείμενο το τροποποιημένο. Συγχαρητήρια στον κύριο Μποβέ. Εγκρίναμε λοιπόν το σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Λοιπόν, το 12 ήδη το κάναμε. Οπότε... Α, Ενημερώνω τους συναδέλφους ότι αποφασίσαμε, συζητήσαμε επανειλημμένα μάλλον το πρόβλημα της χρήσης των κλοβών, των μη τροποποιημένων για τις οροπαραγωγές όρνηθες χρησιμοποιούνται από 1η Πρώτου 2012. Όσον αφορά το πλαίσιο, το πρόβλημα του συντονιστές, συζητήσαμε το ενδεχόμενο προφορικής ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που σας έχει διανεμηθεί. Αν συμφωνείτε, μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτή την προφορική ερώτηση και θα ήθελα να τη βάλουμε στην ημερήσια διάταξη ολομέλεια Ολομέλειας του Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η βούληση των συντονιστών, αλλά βεβαίω αν υπάρχουν σχόλιά σας θα ήθελα να ζητήσετε το λόγο. Δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις, αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Εγκρίνουμε την ε, προφορική ερώτηση. Δεν ζητάει κανείς το λόγο, οπότε πάμε στο σημείο 14 ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στην αγορά ζάχαρης. Κατόπιν ετήματος της ομάδας ΕΛΚ, η Επιτροπή σήμερα θα μας παρουσιάσει την παρούσα κατάσταση της αγοράς ζάχαρης και θα μας δείξει τις ε, συνέπειες της κατάργησης των ποσοστώσεων το 2015. Τι προβλέπετε. Αυτό προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή Verstylen, ε, στον οποίο δίνω αμέσως το λόγο. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Mr. President. Um, let me... Uh, Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι ε, διεξήχθη μια μεταρρύθμιση που αποφασίστηκε το 2005-2006 και άρχισε να εφαρμόζεται το 2006-2007. Βασική αρχή ήταν ότι έπρεπε να προσαρμόσουμε την εσωτερική ε, παραγωγή ως μια προσαρμογή να γίνουμε κατά 85% αυτάρκης και να περιοριστούν οι εισαγωγές. Και έπρεπε να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση αυτή με βάση τις δεσμεύσεις μας για περιορισμό των εισαγωγών εκτός όπλων. Και έπρεπε να τηρήσουμε αυτές τις αρχές. Τώρα, όσον αφορά τις ποσοστώσεις, έχουμε εσωτερική παραγωγή περίπου 14 εκατομμύρια τόνους, ενώ εσωτερική κατανάλωση 16,5 εκατομμύρια. Άρα η διαφορά θα πρέπει να καλυφθεί από εισαγωγές. Παράλληλα με τις ποσοστώσεις ζάχαρης, έχουμε και τη ζάχαρη εκτός ποσοστώσεων, όπου είχαμε στο παρελθόν κάτι άλλο και τώρα μετατράπηκε σε εκτός ποσόστοσης ζάχαρη. Ε, χρησιμοποιείται για βιομηχανική χρήση, τη χημική βιομηχανία, αλλά και για εξαγωγές. Αλλά με μία ποσόστοση 1,305 εκατομμύρια τόνους σύμφωνα με τον ε, ΠΟΕ. Και αν υπάρξει ένα υπόλοιπο, αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί από την ποσόστοση του επόμενου έτους. Έρχομαι τώρα στην κατάσταση της αγοράς. Πάντοτε υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ της κατάστασης στο παρόν έτος σε σχέση με το προηγούμενο. Και θα ήθελα να σας περιγράψω το τι κάναμε το 2010 και το 2011. Αντιμετωπίσαμε μια, ε, μια κατάσταση παγκοσμίως με υψηλές τιμές. Η τιμή δηλαδή της η παγκόσμια τιμή ήταν υψηλότερη σε σχέση με την εσωτερική τιμή. Κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί στο παρελθόν. Και ως συνήθως καλύψαμε το ποσόστοση με 13,5 ε, εκατομμύρια ε, τόνους. Αναμέναμε μια εισαγωγή 2,8 τόνων, εκατομμύριων τόνων και επειδή τα αποθέματα ήταν γύρω στο 1,2 εκατομμύρια, διαπιστώθηκε ότι θα υπήρχε μια έλλειψη στην εσωτερική αγορά. Η Κομισιόν λοιπόν, επειδή είδε την απειλή στρέβλωσης της εσωτερικής αγοράς, έλαβε μέτρα ώστε να υπάρξει επαρκής ποσότητα ζάχαρης στην εσωτερική αγορά και στόχος μας στη διαχείριση αυτής της αγοράς είναι στο τέλος του έτους να έχουμε ένα επίπεδο αποθεμάτων 1,8-1,9 εκατομμύρια τόνους επί τη βάση της εμπειρίας μας του παρελθόντος ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής ροή στην αγορά ζάχαρης. Για να επιτύχουμε αυτό το στόχο κύριε Πρόεδρε, επιτρέψαμε την εισαγωγή επιπρόσθετη των ποσοτήτων ζάχαρης υπό ευνοϊκές συνθήκες 500.000 ε, ε, τόνους ε, και επιπλέον το 50.000. Αλλά μετατρέψαμε και τη ζάχαρη εκτός ποσόστοσης, εντός ποσόστοσης με 5.000 τόνους. Με τα μέτρα αυτά λοιπόν, με καλή ισορροπία μεταξύ εσωτερική σε εσωτερικών αποθεμάτων και εισαγωγών, η κατάσταση τον Οκτώβριο είναι 1,9 εκατομμύρια τόνους σε αποθέματα. Έρχομαι τώρα στο 2011-2012. Επί τη βάση αυτής της παγκοσμίου έλλειψης ε, ποσοτήτων ζάχαρης και των ελλείψεων στην εσωτερική αγορά, μπορούσαν οι παραγωγοί μας να διευρύνουν την παραγωγή τους. Αυτό κατέστη γνωστό πριν από την ε, καλλιέργεια και τούτο είχε ως αποτέλεσμα μια αύξηση ε, κατά 3% των εκτάσεων παραγωγής ζάχαρης. Είχαμε μια πολύ καλή παραγωγή με καλές αποδόσεις και αναμένουμε ε, καλό αποτέλεσμα φέτος. Έτσι λοιπόν καλύπτεται η ποσόστοση, η ζάχαρη σε ποσόστοση και η εκτός ποσόστοσης αναμένεται να είναι 5 εκατομμύρια τόνους. Πέρσι ήταν 8. Υπάρχει δηλαδή μια σημαντική αύξηση της ζάχαρης εκτός ποσόστοσης. Εάν δεν λάβουμε μέτρα, αναμένεται στο τέλος του έτους να έχουμε ένα απόθεμα 1,2 εκατομμύρια τόνους. Άρα λοιπόν λαμβάνουμε μέτρα ώστε να επιτύχουμε το στόχο του 1,9 εκατομμυρίων τόνων, που ήταν και ο στόχος μας. Θα κάνουμε δηλαδή λίγο πολύ το ίδιο που κάναμε και πέρσι. Δηλαδή θα επιτρέψουμε 400.000 τόνους ζάχαρης εκτός ποσόστοσης να μετατραπεί σε ζάχαρη εντός ποσόστοσης και να χρησιμοποιηθεί στην εσωτερική αγορά. Και σύντομα θα ανοίξουμε και μια άλλη δυνατότητα για επιπλέον εισαγωγές μέσω διαγωνισμών. Τούτο σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να εναρμονίσουμε τόσο τις εισαγωγές όσο και την κατάσταση στην εσωτερική αγορά και στις αρχές του προσεχούς έτους θα σκεφτούμε τι επιπρόσθετα μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να επιτύχουμε το στόχο των ε, του 1,9 εκατομμυρίων τόνων στην εσωτερική αγορά. Συνοψίζοντας, κύριε Πρόεδρε, πέρσι λάβαμε μέτρα για να εξισορροπήσουμε την εσωτερική αγορά και βρισκόμαστε στη διαδικασία ε, του να πράξουμε το ίδιο και φέτος ώστε να υπάρξει επαρκής ποσότητα ζάχαρης στην εσωτερική αγορά. Και εδώ σταματώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Διευθύντα. Μπορούμε να ανοίξουμε συζήτηση τώρα. Έχουν ζητήσει να παρεύουν Εράνς Γαρσία, Τζορτζ και άλλοι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε εδώ και έδωσε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα για τον τομέα της ζάχαρης. Όμως κάνατε, λόγο, ε, ή κάνατε λάθος πριν ή κάνετε λάθος τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει απειλή διαγραφής των ποσοστώσεων όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης το 2015. Έχουν περικοπεί σημαντικά οι ποσοστώσεις με την προηγούμενη μεταρρύθμιση. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν υποστεί μείωση 50% στην παραγωγή. Και είναι ελληματική η ευρωπαϊκή παραγωγή. Εισάγουμε ζάχαρη γιατί δεν, μπορώ να κατανοήσω γιατί ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από χρόνια με τέτοιες σημαντικές περικοπές. Η κυρία Φίσερ Μπόλερ για τι σημαντικέ τις σημαντικές αυτές περικοπές της ζάχαρης ε, που ήταν υπεύθυνη διαρωτώ με τώρα Ποιο νόημα έχει με, αυτή την, ε, με αυτά τα ελλείμματα, ποιο νόημα είχε να διαγραφούν, να μειωθούν οι, περι, ποσοστώσεις τότε, να περικοπούν στο παρελθόν και να ε, διαγραφούν πλήρως το 2015. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Οι παραγωγές χώρες πρέπει να έχουν τις ποσοστώσεις μέχρι το 2020. Να έχουμε ευκαιρία να διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή παραγωγή. Να δώσουμε μια ευκαιρία σοβαρή για την παραγωγή μολάσας ε, από πλευρά των ζαχαροπαραγωγών της Ένωσης που έκαναν σημαντική προσπάθεια να προσαρμοστούν στις διαρκείς πιέσεις που υφίστανται και μέσω των μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ ότι στην ΚΑΠ πρέπει να δω στην κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να υπάρξει μια σημαντική αλλαγή όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής και να διατηρηθούν φυσικά οι ποσοστώσεις μέχρι το 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση. Έχω δύο ερωτήσεις. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια είναι τα βασικά δεδομένα ε, και πώς εξηγείται η αύξηση της ε, τιμής ζάχαρης παγκοσμίως. Υπάρχει μείωση παραγωγή, υπάρχει περισσότερη ζήτηση στην Άπο Ανατολή. Ποια είναι τα βασικά αίτια που προκαλούν αυτό το φαινόμενο της αύξησης της τιμής και ποιες είναι και οι προβλέψεις στο μέλλον. Δεύτερον, ένας από τους βασικούς εισαγωγείς ζάχαρης ε, και οι πιλάγιον μου ανέφεραν ότι οι χώρες ΑΚΕ δεν είναι σε θέση να καλύψουν την ποσόστοση που είχαν αναλάβει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο οι χώρες αυτές δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δυνατότητα και σκέφτεστε να, και πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε αυτό, δηλαδή να βγάλετε τις χώρες αυτές εκτός από τα ποσοστώσεις, δεδομένου ότι οι μονάδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν ε, έτσι όπως είχε ε, υπολογιστεί και υπάρχουν πολύ σημαντικές απώλειες. Ο Τζόρτζο Άλμπερτ και μετά Μάρτιν. Ο κύριος Ντές, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως θυμάμαι πολύ καλά οι Γάλλοι συνάδελφοι από τους σοσιαλδημοκράτες ή ε, με εισήγηση που είχαν, εγώ ήμουν σκιώδης εισηγητής για την ε, ομάδα μας και οι άλλοι σκιώδης εισηγητές είχαν συνεισφέρει να αποφύγουμε τα χειρότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε το 2005 να πάει πολύ πιο πέρα με τη μεταρρύθμιση και να μειώσει ακόμα πιο πολύ τις τιμές και το Ευρωκοινοβούλιο παρότι δεν είχαμε συναπόφαση τότε αν δεν είχε αρνηθεί αυτή την εξέλιξη τώρα θα είχαμε πολύ σημαντικότερα ελλείμματα από ό,τι ε, έχουμε και ε, σε σχέση με την ε, πάυση αυτής της καλλιέργειας δεν θα είχαμε δυνατότητα από ευρωπαϊκή παραγωγή να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Τώρα έχει κάνει λάθος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την διαγραφή απάλληψη των ποσοστώσεων το 2015 οι ελλείψεις που υπάρχουν αποκλειστικά οφείλονται στο ότι οι χώρες ΑΚΕ τις ποσώσεις, ποσότητες που μπορούν να δώσουν στην Ευρώπη δεν τις ε, παραδίδουν και έχουμε διαφορές μόνα και αυτό είναι το πρόβλημα για τις ελλείψεις, το έλλειμμα στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι ουσιαστικά υπάρχει αρκετή ζάχαρη διαθέσιμη. Η σημερινή κατάσταση είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης ε, από την ε, βιομηχανία που επεξεργάζεται τη ζάχαρη, μεταποιεί τη ζάχαρη. Και εγώ θεωρώ ότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ε, σωστή πορεία προς την οποία θέλει να πορευτούμε, αν μπορέσει να ε, ακολουθηθεί αυτό το μέτρο θα έχουμε αρκετή ζάχαρη στην Ευρώπη και τώρα για την κοινή οργάνωση αγορά ζάχαρης να καταργηθεί είναι ένα πολύ λαθα, λανθασμένο συμπέρασμα. Σωστά είχε αποφασίσει το Κοινοβούλιο με 90% των ψήφων ότι η μεταρρύθμιση της κοινή οργάνωσης αγοράς θα έπρεπε μέχρι το 2020 να παραταθεί. Εδώ με τη συζήτηση πρέπει να βρεθούμε σε αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν ακολουθεί τη σωστή πορεία. Ευχαριστώ. Bene, grazie Albert Martino. Ευχαριστώ ε, Μάρτιν και μετά ο Ρούμπιξ. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω σε πολλά με τον Άλμπερτ. Πρέπει να δει κανεί την ιστορική κατάσταση και να υπενθυμίσει πώ είχαν τα πράγματα. Στο παρελθόν δεν μπορούσαν αρκετά γρήγορα να ξεκινήσουν τα πράγματα για την πάυση του καθεστώτος ε, του, ε, με την παραγωγή ζάχαρης και τώρα εκείνοι που ζητούσαν ε, να τερματιστεί η ευρωπαϊκή παραγωγή ζάχαρης, ε, τώρα τι θέλουν, θέλουν ε, να λένε ότι είναι ένα εμπόδιο οι ποσοστώσεις και πρέπει να υπάρξει συνέχεια. Είναι κάπως παράλογο αυτό το πλαίσιο συζήτησης και συμφωνώ με τον προλαλήσαντα σε πολλά σημεία οι ποσοστώσεις σε σχέση με την ζαχαροπαραγωγή έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση και 80% καλύπτονται οι ανάγκες από την ευρωπαϊκή παραγωγή. Το θέμα είναι ποια συνέχεια θα δώσουμε. Και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να διατυπώσουμε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το σημείο είναι τόσο στεναρά αντίθετη με τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και δεν προσαρμόστηκε και, δεν, ε, ε, και εδώ πρόκειται και για επιτάχυνση της ε, απάλληψης των ποσοστώσεων τι θα γίνει, μακροπρόθεσμα θα είναι τόσο φθηνή τελικά η ζάχαρη ώστε να υπάρχει αρκετή ποσότητα στην αγορά και να μην υπάρχουν προβλήματα. Πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα ουσιαστικά στο μέλλον. Και αυτό είναι κάτι που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και η υψηλοί δασμοί που εισπράττουμε είναι ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει, πρέπει να παραμείνει έτσι. Τι γίνεται και τι θα γίνει μακροπρόθεσμα με μια πιο ευέλικτη διαμόρφωση του συστήματος ποσοστώσεων. Μήπως θα μπορούσαν να αυξηθούν και οι ποσοστώσεις, να προσαρμοστούμε στις ανάγκες της αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάρτιν Ρούμπιξ και μετά Μισελ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Τι είδου μεταρρύθμιση είναι αυτή τελικά πρέπει να ρωτήσουμε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε ήδη προβλήματα και δυσκολίες και δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας στη ζάχαρη όσο χρειαζόμαστε. Παρότι στην Ευρώπη έχουμε καλά ζαχαρότεφλα που καλλιεργούνται και μπορούμε να παράξουμε αρκετή ποσότητα ζάχαρης. Και κάνουμε λόγο και στη συνέχεια για το ότι η Ευρώπη έχει γίνει εισαγωγέας αντί να είναι εξαγωγέας ζάχαρη, ζάχαρης. Και αυτό δεν είναι κάτι το λογικό και το συνεκτικό, διότι ε, αναπτύχθηκε το σύστημά μας και τελικά αυτό ανταστράφει. Και γι' αυτό θέτω αυτά τα ερωτήματα. Κατανοώ τα πράγματα σωστά ή όχι. Τι είναι εκείνο το οποίο θα συμβεί τώρα που εκτός ποσόστοσης ζάχαρη μεταφέρεται στην εντός, στη ζάχαρη ποσόστοση. Τι σημαίνει αυτό. Λετονοί γεωργοί που θέλουν να ανανεώσουν τις καλλιέργειες ζαχαρότεφλων και την παραγωγή ζάχαρης τελικά από αυτά θα παίρνουν ποσοστώσεις, θα καλύπτονται από αυτές τις ποσοστώσεις ακόμα και όταν δεν προβλέπονται αυτές για τώρα, για αυτό το διάστημα και μετά ακολουθούν οι άλλοι. Εγώ θα ήθελα μία εξήγηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο προηγούμενο κείμενο ε, προβλεπόταν το 2016 να σταματήσει το παλιό σύστημα και τα μέτρα μεταρρύθμισης έπρεπε να αρχίσουν να εφαρμόζονται από το 2015 χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, συζήτηση. Ε, για ποιο λόγο λοιπόν ήρθαμε από το 16 στο 15. Ε, υπάρχει ένας τρόπος σκέψης αβελικός θα έλεγα. Δηλαδή από τη μια διατηρούμε τις ποσοστώσεις στην Ευρώπη και σήμερα ε, δεν μας εξηγούν ε, για ποιο λόγο θα καταργηθεί το όλο σύστημα από το 2015 και εντεύθεν. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον τρόπο σκέψης. Grazie Ευχαριστώ, Μισελ. Ούλρικ και μετά Μαγκίνα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα γίνω δυσάρεστη, φοβούμαι, διότι έχω ένα θέμα αρχή εδώ. Αν στη νέα ΚΑΠ πούμε ότι θέλουμε να σταματήσουμε τις ποσοστώσεις στο γαλακτοκομικό τομέα, αλλά στη ζάχαρη πούμε θα εξακολουθήσουν οι ποσοστώσεις για τη ζάχαρη, αυτό δεν είναι λογικό και συνεκτικό για μένα. Το λέω αυτό προσωπικά, δεν το λέω για την ομάδα μου, προσωπικά το αναφέρω. Όταν ω θέμα αρχή συζητούμε για την κατάργηση ποσοστώσεων και η πλειοψηφία των μελών τη Επιτροπή είναι σε σχέση με το γαλακτοκομικό τομέα να γίνει αυτό, να μην έχουμε ποσοστώσει, ε, δεν έχω δυνατότητα να καταλάβω γιατί στη ζάχαρη θα παραμείνουμε στις ποσοστώσει λέγεται ότι η κατανάλωση ζάχαρης τα τελευταία χρόνια σταθεροποιήθηκε. Έτσι ακούμε. Και η ζάχαρη, λένε, έχει προσαρμοστεί, έχει προσεγγίσει στις τιμές της, τις παγκόσμιες τιμές ε, της ζάχαρης ε. το ίδιο όμως επιχείρημα χρησιμοποιείται και για το γάλα ε, και ότι η τιμή αυξάνεται. Πρέπει να καθαρίσουμε, ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε ποσοστό ισοστέμα αρχής ή όχι. Και αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να μου το εξηγήσει με σωστό τρόπο ώστε να το καταλάβω. Θα ήθελα να μου πείτε προς τα πού κατευθυνόμαστε, προς τα πού πορευόμαστε και ενέκρινα τις προτάσεις Albert Dess για την απάλληψη ποσοστώσεων το 2020. Λέω εδώ ρητά και κατηγορηματικά προσωπικά για μένα δεν γνώριζα τις επιπτώσεις τότε ποιε θα ήταν. Ήταν σημαντικό σε σχέση με το γάλα και το γαλακτοκομικό τομέα στην ΚΑΠ. Πρέπει να αποσαφινιστούν τα πράγματα σε σχέση με την Επιτροπή μας και να υπάρξει ένα αυστηρό πλαίσιο, σαφές πλαίσιο. Δεν είναι δυνατόν τη μια να γίνεται το ένα, την άλλη το άλλο και όλα να αλλάζουν ξαφνικά και να μην ξέρουμε πού πάμε και τι θέλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ούλρικε. Μάριαν και μετά Μπρίτα Ράιμερς. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την Κομισιόν. Θα ήθελα να ρωτήσω. Μιλούμε για την ποσότητα της ζάχαρης, αλλά υπάρχει και θέμα ποιότητας ζάχαρης. Κάποιοι στον τομέα πιστεύουν ότι η ποιότητα, του, η ποιότητα της ευρωπαϊκής ζάχαρης δεν είναι στο επίπεδο που απαιτείται και θέλω μια εξήγηση. Ε, δεύτερον, υποστηρίζω την ερώτηση του Λατωνού συναδέλφου και η Ιρλανδία έχασε ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του κλάδου εξαιτία των μεταρρυθμίσεων. Αλλά ήταν ένα ζωτικό θέμα της, του συστήματος ε, αμύψης φοράς. Ε, και ε, ο κλάδος αυτός έπρεπε να αγωνιστεί για να επιβιώσει, ενώ τώρα πρέπει να αγωνιστούμε για την αναβίωση αυτού του τομέα. Τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν για τις χώρες μέλη να παραγάγουν ας πούμε ζάχαρη για την εσωτερική αγορά ε, καθώς προχωρούμε προς το μέλλον χωρίς το σύστημα των ποσοστώσεων. Ευχαριστώ. Ρίτα Ρέιμερς και μετά Γιάρ παρακαλώ. Αυτό που βλέπω είναι ότι συζητάμε γενικά για τη ζάχαρη. Ουσιαστικά όμως θα έπρεπε να ξέρουμε ότι η ζάχαρη δεν είναι ίδια με τη ζάχαρη. Υπάρχει διαφορά ποιότητας όσον αφορά τα διαφορετικά είδη ζάχαρης. Όλα αυτά όμως τα αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο ισοπεδωτικά όλα τα διαφορετικά είδη. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε μικρή προσφορά σε υψηλής ποιότητας ζάχαρη. Και αυτό οδήγησε στο ότι η χρήστες ε, να μην μπορούν να εξαντλήσουν ε, το ποσοστό, το περιθώριο στην αγορά τους ε, και να αγνοούνται οι ανάγκες των καταναλωτών. Αν δει κανεί τι είδου ζάχαρη αγοραζόταν για να μπορέσει να καλυφθεί η ανάγκη των καταναλωτών στη Γερμανία για παράδειγμα. Και βλέπουμε ότι εδώ αντιδρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν δρά, αλλά αντιδρά. Και σε σχέση με το ε, προτινόμενο σύστημα δεν υπάρχει ένα ευρύ πλαίσιο, αλλά υπάρχει ένα στενό κορσέ, ένα στενό περιοριστικό πλαίσιο σε σχέση με τις, αποθέσεις, ε, με αποφάσεις που δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της αγοράς. Γι' αυτό εγώ είμαι σαφώς υπέρ της ε, κατάργησης των ποσοστώσεων. Θα είμαι σαφώς υπέρ της αποφυγής συστήματος ποσοστώσεων. Δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσουμε θετικά την αγορά. Ούτε πριν από τη μεταρρύθμιση, ούτε μετά τη μεταρρύθμιση. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργήσαν καλά τα πράγματα. Πέρα από αυτό βλέπω με σαφήνεια ότι το δυναμικό διάθεση στην αγορά της ζάχαρης ε, δεν μπορεί να εξαντληθεί, δεν εξαντλείται για να καλυφθούν οι ανάγκες των καταναλωτών. Και όταν έχουμε και ε, το θέμα των εισαγωγών, όταν ε, είναι περιορισμένη η δυνατότητα προσφοράς για κάλυψη των αναγκών και έχουμε θέματα εισαγωγών, αυτά δεν είναι καλά για την αγορά και πρέπει να αναγνωρίσουμε επιπλέον ότι οι συνήθειες οι διατροφικές αλλάζουν στον κόσμο παγκόσμια και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Υπάρχει άνοδος του επίπεδου ευημερίας σε πολλές χώρες και αλλαγή διατροφικών συνηθιών και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση με τις ανάγκες κάλυψης των, ε, της ζήτησης των καταναλωτών με ζάχαρη. Για να ικανοποιηθούν αυτές οι τάσεις πρέπει εδώ να ακολουθήσουμε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ε, προσαρμογής ε, για να ικανοποιηθούν αυτές οι καταναλωτικές ανάγκες. Πρέπει να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις, απο, τις ποσοστώσεις, να καταργήσουμε τις ποσοστώσεις. Το ότι είναι κάτι το οποίο πλήττει πολλούς ή τους εκπλήττει το ότι το 2014 πρέπει να υπάρξουν ε, αλλαγές. Αν διαρκώς αλλάζουν οι παράμετροι, έχει δίκιο η συνάδελφος ότι τα πράγματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν καλά. Ευχαριστώ Μπρίτα. Γιάρ και μετά τα ραμπέλα επόμενη. Ναι, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν μια προσωπική άποψη πρώτα και μετά μια γενική πολιτική παρατήρηση και μετά σύντομες ερωτήσεις. Προσωπική άποψη. Στην Ανατολική Γερμανία έχουμε πρόβλημα σε σχέση με τους, ε, τις καταναλωτικές ανάγκες είτε ήταν ε, σε ποσόστοση ή εκτός ε, ουσιαστικά έχουμε τις δομές του σοσιαλιστικού καθεστώτος που από τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας καθοριζόντουσαν. Αν ρωτήσετε τους γεωργούς αν κατανέμονται δίκαια τα ποσοστά ζαχαρότευτλων σας λένε όχι διότι προηγούμενα είχαμε και το κομμουνιστικό καθεστώς και έχουμε ένα περιφερειακό πρόβλημα και γενικά υπάρχει συνένεση όταν έχουμε τεχνητές ποσοστώσεις που θέλουμε να τις καταργήσουμε και υπάρχει συνένεση γι' αυτό τώρα η πολιτική παρατήρηση κύριε Ρόντος πρέπει να είμαστε ειλικρινείς κανονικά έχουμε γεωργικά μία άλλη πορεία που ακολουθείται σε σχέση με τις ποσοστώσεις. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, τώρα έχουμε στο παρόλα αυτά, έχουμε καεί από την εμπειρία του παρελθόντος. Είμαστε και, έχουμε μάθει πλέον ε, και γι' αυτό δεν τα καταφέραμε σωστά και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν ήταν ομαλή η προσγείωση. Ήταν μάλιστα απότομη και ανώμαλη προσγείωση. Γι' αυτό πρέπει στη ζάχαρη να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί καλύτερα θα ήταν να καταργηθούν οι ποσοστώσεις και κανένας ε, να μην το αντιληφθεί, δηλαδή εννοώ με το κανένας για τους καταναλωτές. Και τώρα έχει τη ερώτηση προς την Επιτροπή. Δημιουργείται ανασφάλεια. Δεν θέλουμε άλλη μια ανώμαλη προσγείωση. Γι' αυτό η ερώτησή μου τώρα την έθεσε και ε, ε, προλαλή σας. Τι, προ, ποιες προγνώσεις υπάρχουν, πόσο ασφαλής είναι οι προγνώσεις τιμών ε, από πλευρά σας για υψηλό επίπεδο τιμών και το τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να είναι απλό το σενάριο αλλά δεν είναι απλό στην εφαρμογή και εύκολο και υπάρχουν ίσως προβλήματα όταν δεν είναι ευδοκιμή. Τώρα τίθεται το ερώτημα, ποιο περιθώριο υπάρχει, περιθώριο λιγμών στο σύστημα μέσα στις ποσοστώσεις, ώστε να ρυθμίσουμε τις ποσότητες παραγωγής. Την ποσόστοση γάμα, C, μπορούμε χωρίς πρόβλημα να την ε, διαθέσουμε στην Ευρώπη αν, είναι, αν υπάρχει ζήτηση ίσως. Τέτοιου είδους ερωτήσεις που πρέπει να ανήκουν στο πακέτο μέτρων εμπιστοσύνης. Αυτά χρειάζονται οι γεωργοί μας. Διότι αν λειτουργήσουν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αν υπάρξει με τις αλλαγές ε, μια δυνατότητα εμπιστοσύνης, θα μπορούσαμε χωρίς προβλήματα, χωρίς τριβές, στο μέλλον να καταργήσουμε τις ποσοστώσεις. Τότε θα είχαμε μια κατάσταση win-win. Αλλά Πρέπει γενικά να αναγνωρίσουμε πολιτικά ότι εμείς ουσιαστικά βρισκόμαστε καθοδόν το ε, σύστημα των ποσοστώσεων να ε, το αντιμετωπίσουμε καταργώντας το ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιά. Μαρκ Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ε, θα ήθελα να μην εισαγάγουμε την πολιτική στην αγορά. Η αγορά έχει τους δικούς της κανόνες ε, και δεν θα πρέπει να υιοθετήσουμε υπερβολικά φιλελεύθερες θέσεις όπως καμιά φορά η Κομισιόν. Αυτό που χρειάζεται ενδεχομένω είναι μια πολιτική ρύθμιση της παραγωγής ούτως ώστε να είναι πιο εύκαμπτη και να μπορεί να ανταποκρίνεται στην αγορά να προσαρμόζεται στην αγορά αλλά και σε περιόδους ε, κρίσης. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και πρόκειται για μια γενική αρχή ότι το, είχαμε αποφασίσει ότι το 2005 θα διατηρήσουμε την παραγωγή ε, στο νότιο τμήμα, ενώ το, όλο το βόρειο τμήμα από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία κλπ. θα έπρεπε να εξαλειφθεί. Και βεβαίως αυτό προκαλεί την αντίδραση των παραγωγών και του κλάδου, διότι απαιτεί ε, αποζημιώσεις για ποιο λόγο για να αναδιαρθρωθεί ή να μετακομίσει σε άλλες υπήρους. Και τώρα είμαστε αναγκασμένοι να εισαγάγουμε ζάχαρη. Ξεκάθαρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να σκεφτούμε να έχουμε μια πολιτική ρύθμιση βεβαίως με ευελιξία ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις αγορές. Και αυτό ισχύει για τη γεωργία αλλά και για την ε, βιομηχανία. Όλος ο κόσμος είναι ανοιχτός. Η Κίνα, η ε, Βραζιλία, οι πάντες, εκτός από την Ευρώπη η οποία κλείνει τις πόρτες στη βιομηχανία, στη γεωργία, στη στη βαριά βιομηχανία κλπ. Ενώ οι άλλοι ανοίγουν τις αγορές. Και εμείς και εγώ θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό στην Επιτροπή Ίνκο για την εσωτερική αγορά. Και εμείς ανοίγουμε τις πόρτες προς όλους και ουσιαστικά ξυλώνουμε το δικό μας οικοδόμημα το έναντι όλων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο ευέλικτοι με την απαραίτητη βεβαίως ρύθμιση η οποία είναι απολύτως απαραίτητη δεν πρέπει να καταργήσουμε εντελώς τις ποσοστώσεις όπως κάναμε στον τομέα του γάλακτος διότι πριν από 20-25 χρόνια δεν είχαμε αυτές τις φοβερές κρίσεις όπως είχαμε πρόσφατα, όπως το 2009 παραδείγματος χάρη, διότι είδαμε τι ακριβώς συνέβη. Οι τιμές αυξήθηκαν ε, διπλασιάστηκαν ουσιαστικά. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια ρύθμιση ανάλογα όμως με τις ανάγκες της αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Μάρτιν Όστριγκερ για λίγο και μετά θα ακολουθήσουν άλλοι. Συγγνώμη που ζήτησα και πάλι τον λόγο, αλλά η συζήτηση για τις προσωστώσεις βρίσκω ότι είναι ενδιαφέρον βέβαια ότι εκείνοι που υπάρχουν από τη μία μεριά λένε ότι είναι για την κατάργηση των ποσοστώσεων, οι άλλοι είναι υπέρ της διατήρησή του. Σε πολλά σημεία ωστόσο πρέπει να διαφοροποιούμε τα πράγματα. Το ένα δεν ταιριάζει πάντα με το άλλο. Και έχουμε και τη συζήτηση για το κρασί. Όλα να απορριθμιστούν. Τι θα γίνει στο τέλος. Και αν όλα απορριθμιστούν και απελευθερωθούν, είναι σαφές πρέπει να, να ε, διαφοροποιήσουμε τι θα κάνουμε σε σχέση με τις, ε, τη διαχείριση των ποσοστώσεων και εναλλακτικέ λύσεις. Λοιπόν, η ερώτησή μου θα ήταν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα έχει εγκρίνει ένα γλυκαντικό το Σέβια που στην ε, ποτοβιομηχανία και στη ζαχαροβιομηχανία διαδραματίζει ένα ρόλο. Ποιες επιπτώσεις θα έχει στην αγορά λευκής ζάχαρης αυτός, αυτή η γλυκαντική ουσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τη Μαρέη Μακίνε και τον συνάδελφο από την Λετωνία. Ναι, θέλετε να παραγάγετε ζάχαρη, αλλά υποδομές υπάρχουν. Αυτό δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τους γεωργού. Υπάρχει και η διαδικασία. Και οι άνθρωποι πρέπει να είναι απόλυτα βέβαιοι ότι ε, θα κατασκευάσουν ας πούμε μια μονάδα η οποία θα λειτουργήσει για αρκετά χρόνια και έτσι θα διαθέσουν τα χρήματά τους. Προ την Κομισιόν τώρα. Έχετε κάνει μια αξιολόγηση επιπτώσεων για το τι ακριβώ συμβαίνει. Διότι το ζαχαρό τεφτλό είναι ένα είδο το οποίο παράγεται σε πάρα πολλές χώρες. Πέρσι Πέρσι έχασα το 1 τρίτο της παραγωγής εξαιτία του πολύ ψυχρού μόνα και καταλήξαμε 16 τόνους κατά ε, μονάδα. Φέτος θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση, θα είναι 13 τόνους. Αν λοιπόν καταργήσουμε τις ποσοστώσεις και πούμε ότι είναι ελεύθερα τα πάντα για όλους, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι καλλιέργειες θα στραφούν στις περιοχές εκείνες όπου έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια παραγωγής. Ανατολική Γαλλία, ε, νότιες χώρες κλπ. όπου οι ε, χειμώνες είναι πολύ πιο ήπιοι. Δηλαδή αυτό το σκεφτήκατε λίγο πιο μπροστά, προβλέπετε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Ευχαριστώ όλους σας. Δίνω το λόγο και πάλι στον Διευθυντή Βεστάιλερ και εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τις ανησυχίες των συναδέλφων. Πριν διαλυθούν όλα αυτά τα μέσα διαχείρισης της αγοράς, προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα ισχυρό προστατευτικό δίκτυο μέσα διαχείρισης των κρίσεων ε, διαφορετικά κινδυνεύουμε να κάνουμε επιλογές που μπορούμε, μπορεί να μετανιώσουμε αργότερα. Λοιπόν και διευθυντά έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα προσπαθήσω να απαντήσω στις διάφορες ερωτήσεις αρχίζοντας ε, με την απάντηση προς τον κύριο Γκαρσία, ο οποίος εξέφρασε την λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχει μια, ένα έλλειμμα στην εσωτερική αγορά. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι όπως είπα και στην εισαγωγική μου παρέμβαση αυτό ήταν αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης που ελήφθη το 2005-2006 και είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι έχουμε διεθνείς, διε, διεθνείς ε, δεσμεύσεις ε, και πιο συγκεκριμένα αυτή των ε, ε, την οποία συμφωνήσαμε εκτός των όπλων. Άρα λοιπόν ε, οι ποσοστώσεις είναι συγκεκριμένες και η εισαγωγή δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια τόνους. Έπρεπε λοιπόν να σχεδιάσουμε ένα σύστημα το οποίο θα έπρεπε να λάβει υπόψη και τις εισαγωγές, όπως εξήγησα νωρίτερα. Μια άλλη ερώτηση αφορούσε στην ε, τιμή σε παγκόσμια, στην παγκόσμια αγορά και την εσωτερική αγορά. Ε, Εξαιτία λοιπόν των μεταρρυθμίσεων που υιοθετήσαμε έπρεπε να μειώσουμε την τιμή της εσωτερικής αγοράς. Έπρεπε λοιπόν να προσαρμοστούμε στις παγκόσμιες τιμές. Έπρεπε να καθορίσουμε μια τιμή αναφοράς γύρω στα 400 ε, ευρώ ανατόνο. Και τα επόμενα χρόνια υπήρξε μία σύγκριση μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών τιμών και τούτο οφειλόταν στην διαθεσιμότητα στην εξωτερική αγορά και την εσωτερική. Ε, και κάποια στιγμή, πέρσι μάλλον, αυξήθηκαν οι τιμές της εξωτερικής αγοράς και αυτό ήταν μία αναμενόμενο. Έχουμε τώρα μια πολύ καλύτερη συγκομιδή σε 172 εκατομμύρια τόνους. Οι τιμές πέφτουν και πάλι και παρατηρούμε επίσης μια διαφορά μεταξύ της, ε, της τιμής στην εσωτερική αγορά και στην εξωτερική αγορά. Και υπάρχει ένα χάσμα, το οποίο όμως δεν είναι δεδομένο και για το μέλλον. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη στο πλαίσιο της πρότασής μας κατάργησης των ποσοστώσεων ή μη ανανέωση του καθεστώτος ποσοστώσεων μετά το 2015. Διαπιστώσαμε μια πραγματική ε, σύγκληση ε, στο επίπεδο τιμών στην εσωτερική και την εξωτερική αγορά. Και τούτο όχι μόνο προς το επίπεδο των τιμών. Επίσης και το κόστος παραγωγής μας, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην όλη συζήτηση, μειώθηκε, διότι οι αποδόσεις ανά εκτάρια βρίσκονται σε σταθερή αύξηση. Άρα λοιπόν προσεγγίζουμε ένα κόστος παραγωγής που βρίσκεται πολύ κοντά στην παγκόσμια, στο παγκόσμιο επίπεδο. Θα μπορέσουμε λοιπόν να ανταγωνιστούμε με την παγκόσμια ε, παραγωγή ζάχαρης και το κόστος αυτής. Συνεπώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκυριακή κατάσταση θα έλεγα τόσο ως προς τις τιμές όσο και ως προς το κόστος παραγωγής που θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε ένα σύστημα χωρίς ποσοστώσεις. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω επίσης τους ενδιαφερόμενους ότι αυτή τη στιγμή η Κομισιόν διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της εσωτερικής αγοράς, αλλά υπάρχουν περιορισμοί στις εξαγωγές μπορούμε να εξαγάγουμε μόνο 1,3 εκατομμύρια τόνους ζάχαρη εκτός ποσόστησης στο πλαίσιο των διεθνών μας συμφωνιών. Και αν καταργηθούν οι ποσοστώσεις, οι εσωτερική παραγωγή θα μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες στην εσωτερική αγορά αλλά και την εξωτερική. Τώρα, στο πλαίσιο των προτάσεών μας μετά το 2013 έγινε ένα γενικό σχόλιο μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων. Έρχομαι τώρα σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ετέθη το ερώτημα για ένα νέο προϊόν, το στέβια, που είναι ένα γλυκαντικό. Δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορέσει να αντικαταστήσει τη ζάχαρη. Ε, ε υπάρχουν πολλά τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν σχετικά με αυτά τα γλυκαντικά, την ασπαρτάμι κλπ. Και αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει τις τιμές της ζάχαρης. Μία άλλη ερώτηση σχετικά με τους δασμούς. Όχι, δεν έχουμε δασμούς. Έχουμε δασμούς όμως σε κάποιες ποσοστώσεις. Ανάλογα με την κατάσταση στην αγορά μπορούμε να τα προσαρμόσουμε. Άλλη ερώτηση. Δεν μπορούμε εν τω μεταξύ να αυξήσουμε τις ποσοστώσεις. Για... Και πάλι. Κύριε Πρόεδρε, προχωρήσαμε στη μεταρρύθμιση και ο Ευρωπαίος καταναλωτής πλήρωσε όπως γνωρίζετε για τη μεταρρύθμιση και πλήρωσε και για την αναδιάρθρωση όταν δηλαδή καταργήσαμε τις ποσοστώσεις στην αγορά. Και δεν είναι λογικό και πάλι να εισαγάγουμε την ποσόστοση. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Και να υπενθυμίσω ότι η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα όταν υπάρχει απειλή διαταραχής της εσωτερικής αγοράς να περάσει την, την ε, ζάχαρη εκτός ποσόστοσης, την ε, ζάχαρη εντός ποσόστοσης, ούτως ώστε να προσαρμοστεί στις ισχύουσες, στην ισχύουσα κατάσταση, στην ισχύουσα στην αγορά κατάσταση. Έτσι απαντώ και στο ερώτημα ε, εάν πρόκειται να εισαγάγουμε επιπρόσθετες ποσοστώσεις. Ε, μετά τέθη το ερώτημα γιατί καταργούμε τις ποσοστώσεις στα γαλακτοκομικά και όχι στη ζάχαρη. Κοιτάξτε, υπήρχε μια γενικότερη τάση να καταργηθούν οι ποσοστώσεις και οι περιορισμοί στην παραγωγή. Αρχίσαμε τις μεταρρυθμίσεις από το 1992 θα έλεγα και για να προσανατολιζόμαστε προς την αγορά και το ένα εκτεταμένο σύστημα ποσοστώσεων δεν συντεριάζει με αυτή την προσέγγιση. Γινόμαστε όλο και περισσότερο παγκόσμιος εταίρος. Άρα δεν πρέπει να επιβάλλουμε περιορισμούς στους παραγωγούς μας για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε ελεύθερα σε αυτές τις διεθνείς εξελίξεις. Μια άλλη ερώτηση αφορούσε στην κατάσταση στην Ιρλανδία. Είχαμε ένα σύστημα όπου κάθε χώρα μέλος και κάθε εταιρεία μπορούσε να λάβει την απόφαση αν θα συνέχιζε να λειτουργεί στο πλαίσιο ε, του συστήματος χαμηλών τιμών can they uh, survive Έπρεπε λοιπόν κάθε εταιρεία να αποφασίσει αν θα προσαρμοζόταν στη νέα κατάσταση τιμών ή όχι. Ή αν θα έπρεπε να σταματήσει τη λειτουργία και να διαλυθεί. Και στην περίπτωση αυτή βεβαίως υπήρχε η ανάλογη αποζημίωση. Άρα λοιπόν ε, δεν υπάρχει περίπτωση να επανεισαγάγουμε ποσοστώσεις στις χώρες εκείνες οι οποίες έλαβαν αυτή την απόφαση. Έγιναν επίσης και κάποια σχόλια με την έννοια σε ποιο βαθμό μπορούμε να προσαρμόσουμε το σύστημα ποσοστώσεων και πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία κλπ. Ε, κύριε Πρόεδρε, το 2015 θα έχουμε επαρκή μέσα εργαλεία στην διάθεσή μας και την απαραίτητη ευελιξία για να προσαρμοστούμε στις νέες καταστάσεις. Και ταυτόχρονα θα υπάρχει και επαρκής ποσότητα ζάχαρη στην εσωτερική αγορά. Για μία ακόμα φορά ετέθε το ερώτημα περί των τιμών. Ε, θα μας επιτρέψει η κατάσταση των τιμών να καταργήσουμε τις ποσοστώσεις εντελώς. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια σύγκληση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών τιμών και ότι και το κόστος παραγωγής μας έρχεται πιο κοντά ή έφτασε το παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, ως προς το μέλλον, μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων, διαπιστώνουμε ότι ε, ότι προσαρμόστηκε το κόστος παραγωγής από ζαχαροτάθλα. Ε, βεβαίως ε, η παραγωγή θα συνεχίζεται στις περιοχές εκείνες όπου υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα αποδόσεων, ε, δυνατότητα μεγαλύτερων αποδόσεων και εδώ πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε μέσα σε μια κατάσταση παγκόσμιας αγοράς. Καλώ δεν ξέρω αν ικανοποιήθηκαν όλοι από τι εξηγήσει που μα έδωσε ο κύριο ε, Διευθυντή. Όμω ε, έγινε μια ευρεία συζήτηση επί ενό θέματο, επί του οποίου σίγουρα θα επιστρέψουμε στι συζητήσει που αφορούν τη μεταρρύθμιση τη αγροτική πολιτική. Πάμε στο τελευταίο σημείο, το 15, πληροφορίε από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τι προετοιμασίες για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομία, παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της ε, γεωργία. Όπως ε, ξεκινά από τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, είναι απαραίτητη η καινοτομία. Προετοιμαστεί για το μέλλον η γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια σύμπραξη λοιπόν για την καινοτομία με στόχο την προώθηση έναν αποδοτικό, έναν ε, αποτελεσματικό ε, αγροτικό τομέα που θα είναι αποδοτικός με χαμηλές εκπομπές. Αυτή η σύμπραξη ε, καλεί τους εταίρους ενδιαφερόμενους να διευκολύνουν την εφαρμογή της ενοτομίας και της έρευνας σε συγκεκριμένες δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας μιλήσει λοιπόν για αυτό το πρόγραμμα, για σημαντικό, το σημαντικό πρόγραμμα δίνοντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον εκπρόσωπο που πρέπει να είναι ο κύριος Σιλ της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργίας. Πάρε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προσέγγιση της εταιρική σχέσης για την καινοτομία προέρχεται από την πρωτοβουλία Ναυαρχίδα για την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη υπάρχει αναφορά σε αυτή την εταιρική σχέση ε, καινοτομίας για τη γεωργία. Αλλά μετακινούμαστε αμέσως επί του θέματος ουσίας και στους στόχους, ξεκινώντας από τις προκλήσεις έχουμε μια πρόγνωση 70% αύξησης όσον αφορά την αγορά στο μέλλον και ήδη έχουμε θέματα ανταγωνισμού λόγω και της αυξανόμενης ζήτησης βιομάζας ε, ενεργειακών προϊόντων και της διασφάλισης βιοπικιλότητας μέσω των μέτρων και είναι απόλυτα σαφές σε μια τέτοια κατάσταση έχοντας αυξανόμενη ζήτηση αυτό θα οδηγήσει σε μια αντίδραση που θα υπάρξει από τον τομέα της γεωργίας. Πάντα ενθυμούμενοι ότι στο παρελθόν αύξηση παραγωγικότητας και είχαμε ιστορία επιτυχιών που ήταν έτοιμοι οι γεωργοί στο παρελθόν να ανταποκριθούν στις πρόσθετες ανάγκες. Και είδαμε ότι εν μέρη επετέφθησαν οι στόχοι εις βάρος του περιβάλλοντος και εις βάρος των φυσικών πόρων. Από αυτά μπορούμε να συναγάγουμε το συμπέρασμα βίαστα ότι αν η γεωργία απλώς αντιδρά στην αυξανόμενη ζήτηση με βάση τις προηγούμενες, ε, τα προηγούμενα πρότυπα θα έχουμε σημαντικά προβλήματα με τους υδάτινους πόρους, με το έδαφος, ε, με την ε, βιοπικιλότητα και όλα αυτά πρέπει να τεθούν εν τάξη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η αύξηση της παραγωγής. Ναι, υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για τη ζήτηση, αλλά πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή ευθυγραμμιζόμενη πάντα με μια αϊφόρο προσπάθεια όσον αφορά τη διαχείριση και διαχειρισιμότητα των ε, ε, πόρων, φυσικών πόρων. Και αυτό απαιτεί όχι μόνο δράση στον πρωτογενή τομέα, διότι σε πολλές πτυχές λύσεις και ε, στόχοι μπορούν να επιτευχθούν και πριν και πιο κάτω από την εφαρμογή ε, προηγούμενων μέτρων. Και έχουμε και το θέμα του 25% όσον αφορά την ε, παραγωγή τροφίμων. Και αν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες, μπορούμε να ανακουφίσουμε τη μεγάλη πίεση στον πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά όμως είναι λύσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των μελλοντικών προκλήσεων και αντιμετώπισης ε, ε, των προβλημάτων που πρέπει να επιλύσουμε Πρέπει να δούμε ποιες μεθόδους έχουμε στη διάθεσή μας, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στην ανάπτυξη και να διασφαλίσουμε ότι αυτή η έρευνα θα μπορέσει να οδηγήσει σε καινοτόμες δράσεις που θα είναι στη διάθεση των γεωργών επιτόπου και θα είναι αποτελεσματικές. Τούτων λεχθέντων υπάρχει πολύ καλή έρευνα και ποιότητα στην έρευνα όπως διεξάγεται σήμερα και πρέπει πολλές φορές να δούμε ότι πρέπει να ακολουθηθεί η καινοτόμος προσέγγιση στην πρακτική εφαρμογή. Απ' την άλλη πλευρά, γεωργοί θέλουν να προσαρμόσουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις προκλήσεις, όμως ακούμε συχνά παράπονα ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι σωστά προσαρμοσμένα και σχεδιασμένα για τις δικές τους ανάγκες και είναι δύσκολο οι γεωργοί να δουν πώς οι ανάγκες τους μπορούν να διευθετηθούν από την ε, έρευνα όπως διεξάγεται σήμερα. Τούτων λεχθέντων πρέπει τα πρακτικά αποτελέσματα λοιπόν της έρευνας να εφαρμοστούν στην πρακτική. Αυτό χρειάζεται, για να γίνει αυτό χρειάζεται ε, η δράση συμβούλων και ε, προσαρμογή. Πρέπει να προσαρμοστεί η προσέγγιση της έρευνας λαμβάνοντας υπόψη όλη την αλυσίδα στην παραγωγή και όχι μόνο το πρωτογενές σκέλος. Και πρέπει ιδιαίτερα να διασυνδεθούν όλα, τα, όλοι οι ενδιάμεση κρίκοι στην παραγωγή, διότι υπάρχουν πολλές δράσεις που μπορούν να παράξουν αποτελέσματα. Όμως δεν διασυνδέονται επαρκώς μεταξύ τους σε ένα συνολικό πλαίσιο, σφαιρικά, ώστε να μπορέσουν οι προσπάθειες να στοχοθετηθούν σε ένα σωστό κοινό αποτέλεσμα. Γι' αυτό συμπέρασμά μας πρέπει πολλά περισσότερα να γίνουν στη διαδικτύωση και αλληλοσύνδεση να μπορέσουν αυτά τα υφιστάμενα μέτρα να αλληλοσυνδεθούν ώστε να υπάρξει συνέργεια, συμπληρωματικότητα, παραπληρωματικότητα. Καταλήγω στα μέτρα για τα μέτρα τα οποία σε σχέση με την ε, ανάπτυξη δράσεων μέσα στο πλαίσιο της ΚΑΠ και της μεταρρύθμισής τους, τη μεταρρύθμισής της για να ε, αριθμίσω κάποια υπάρχει δυνατότητα σύμβουλοι, επιστήμονες, γεωργοί μη κυβερνητικέ οργανώσεις επιτόπου να συνέρχονται για να αντιμετωπίσουν ένα χειροπιαστό πρόβλημα που υπάρχει σε μια για παράδειγμα γεωργική εκμετάλλευση. Μεταφορά τεχνογνωσίας και γνώσης μέσω συμβούλων και υπηρεσιών συμβουλευτική, ώστε να υπάρξει επένδυση και υποστήριξη επενδύσεων και υποστήριξη μέτρων φιλοπεριβαλλοντικών για παράδειγμα ή τοπική ανάπτυξη, που θα επιτρέψουν όλα αυτά σε μια δικτύωση να έχουμε μια εργαλειοθήκη, ένα σύνολο μέσων στα χέρια μας που θα μπορέσουν να ε, επιτύχουν ένα στόχο από κοινού καλύτερα από ότι αν είμαστε κατακαιρματισμένοι για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και προτιθέμεθα να ε, συνδέσουμε ένα δίκτυο, εξειδικευμένο δίκτυο για την εταιρική σχέση για την καινοτομία που θα διασφαλίζει την σωστή και αποτελεσματική ροή πληροφοριών προς τους εταίρους, θα δίνει τις πληροφορίες για τις ευκαιρίες για την έρευνα και την ανάπτυξη σε σχέση με τη γεωργία θα συνδέει τους γεωργούς ώστε να υπάρχει ανταλλαγή βέλτιστων ε, πρακτικών ε, από πλευράς εμπειριών και τεχνικών και φυσικά θα διασφαλιστεί μια συστηματική αμφίδρομη δράση, feedback, ε, όσον αφορά τις ανάγκες τους ε, και τα αποτελέσματα και την διεξαγωγή έρευνας ώστε να μπορέσουν τα μέτρα αυτά να είναι τα καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Για την έρευνα τώρα υπάρχει ένας ε, ο χρονορίζοντας του μέχρι το 2020 και βρίσκονται καθοδόν ε, υπό εκπόνηση τα μέτρα για αυτόν τον, την επίτευξη αυτού του στόχου. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε και πώς θα τα πετύχουμε αυτά σε σχέση με τις προσεγγίσεις μας. Η, τα σχέδια ευρωδικτύου Euronet για το έδαφος ε, και τους υδάτινους πόρους, πλατφόρμες τεχνολογίας. Δεν είναι ένα θέμα επικάλυψης ή ε, μίμησης και διπλασιασμού προσπαθειών. Είναι ανάγκη διασύνδεσης ε, των μέτρων και των δράσεων και δραστηριοτήτων ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα συνέργειας. Τώρα, για την ίδια την ιδέα της καινοτόμου εταιρικής σχέσης θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να ανταποκριθεί σε σχέση με τις ανάγκες μόνο η δράση εκ των άνω προς τα κάτω. Όχι, πρέπει η προσέγγιση να είναι εκ των κάτω προς τα άνω. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις τεχνικές ανάγκες, τις ανάγκες που υπάρχουν στο επίπεδο των μονάδων εκμετάλλευσης, γεωργικών μονάδων εκμετάλλευσης. Εδώ υπάρχουν θέματα τεχνολογίας, διαφάνειας, τον τρόπο με τον οποίο η επιμελητιακή υποστήριξη θα διασφαλιστεί και στο τέλος η τροφική αλυσίδα, η επιστική αλυσίδα μέχρι το τελικό καταναλωτή από το πεδίο της παραγωγής από το χωράφι στο πιάτο. Όλα αυτά αφορούν την ε, καινοτόμο εταιρική δράση. Βλέπουμε ότι οι εξελίξεις ε, θα πρέπει υπό αυτό το πρίσμα να εξεταστούν στην προσέγγισή μας. Έχουμε εγγράψει θέματα στην καινοτόμο εταιρική σχέση για την ε, ανάπτυξη αυτής της νέας προσέγγισης συν επιπλέον τις προτάσεις ε, για, την, για ένα δίκτυο καινοτόμο εταιρικής ε, σύμπραξης. Επιπλέον όσον αφορά την γεφυροποίηση, δημιουργία γεφυρών όσον αφορά την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή, επικοινωνία και διάχυση στοιχείων και προς το Κοινοβούλιο. Η επίσημη καθέλκυση αυτής της εταιρική σχέσης θα ξεκινήσει μετά την ευνοϊκή γνωμοδότηση, την έγκριση από πλευράς Κοινοβουλίου όλων αυτών των προθέσεων. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί αυτό το μέσο διευκόλυνσης. Ε, το καλύτερο δυνατό θα ήταν το 2012. Αυτό θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να επικεντρωθούμε στην εξέταση εξέταση της επόμενης προγραμματικής περίοδου, ώστε να μην υπάρχει μια κατακαιρματισμένη ή ξαφνική, ας το πω έτσι, ε, εκκίνηση που δεν θα έχει λάβει υπόψη μια επαρκή συζήτηση των πραγμάτων που θα πρέπει να έχουν υποσυζήτηση οριμάσει για να λειτουργήσουν σωστά. Έτσι πρέπει να προσεγγίσουμε την υλοποίηση της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου υπό αυτό το σφαιρικό πρίσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σίλε. Ξεκινάει η συζήτηση. Κάποιοι συνάδελφοι να μιλήσουν. Πρώτα κύριε Μαγκίνε, Ντόρφμαν και Ρέιμερ είναι οι επόμενοι. Έχει το λόγο, Μάριον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την Επιτροπή για την παρουσίαση. Το θέμα αυτό συζητείται στις χώρες μέλη. Και πραγματικά ακόμα δεν μπορεί κανείς να δει την ουσία. Δηλαδή, το, το περιεχόμενο πάνω στο σκελετό της ιδέας. Δηλαδή, απαιτείται περισσότερη έρευνα και μεταφορά γνώσεων. Τώρα, σχετικά με κάποια πιο συγκεκριμένα σημεία. Στη νέα κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2020, αυτή η ιδέα είναι μέρος της πρότασης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Υπάρχει όμως πρόβλεψη και, πο... και πώς θα συμβεί αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Αντιλαμβάνομαι ότι καθυστερεί κάπως η πρόταση επειδή θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα από τα πιλωτικά προγράμματα. σχετικά με την ενεργό γύρανση και θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Και επίσης σε διάφορες χώρες μέλη οι υπηρεσίε έρευνα αλλά και παροχή συμβουλών είναι εντελώς ε, διαφορετικές. Κάποιες είναι ιδιωτικέ, άλλε χρηματοδοτούνται από το κράτος. Πώ θα αντιμετωπιστεί αυτή η μεικτή κατάσταση στις χώρε μέλη. Και το τελευταίο σχόλιο, το θέμα της ε, βιωσιμότητα. Συμφωνούμε, θέλουμε και οικονομική βιωσιμότητα στη Γεωργία, παράλληλα με την περιβαλλοντική δηλαδή. Και εικάζω ότι και τούτο θα αποτελέσει μέρος αυτής της πρωτοβουλίας. Δηλαδή πώς οι αγρότες θα εξασφαλίσουν ένα εισόδημα με βάση τις απαιτήσεις που έχουμε με ε, παραγωγή τροφίμων ε, υψηλής ποιότητας, ε, με διακυμάνσεις στις τιμές, αλλά ταυτόχρονα τίθεται να αμφιβόλω η οικονομική βιωσιμότητα μιας τέτοιας δραστηριότητας. Ευχαριστώ. Ο Χέρμπερτ, μετά η Μπρίτα. Ο Χέρμπερτ, ευχαριστώ πρόεδρε. Με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες ε, σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ. Πιστεύω ότι οι προκλήσεις ταυτόχρονα για την αηφορία και εντατικότερα να παράγουμε είναι μια κεντρική κέρια, κομβική πρόκληση των επόμενων ετών και δεκαετιών για τη γεωργία. Αν θέλουμε την παγκόσμια ζήτηση σε τρόφιμα να την καλύψουμε ως ανάγκη. Και θα έλεγα επίσης Έχουμε και την πρόταση για μια μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ και να δούμε ότι στον δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να προβλέπονται κονδύλια, αλλά για όλα αυτά δεν θα επαρκούν και είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα και έχουμε ξεχάσει πλήρως φαίνεται αυτό το θέμα για τη χρηματοδότηση. Αν δούμε τα προτινόμενα μέτρα για, την πρώτο, για τον πρώτο πυλώνα και την αγρανάπαυση και πώς αυτό συσχετίζεται με την εντατο, εν, εντατικοποίηση και την αηφορία δεν μπορώ να κατανοήσω πώς συνδέεται. Πρέπει να δούμε ότι έχουμε στόχους αλλά που πολύ δύσκολο μπορεί να επιτευθούν όταν ακολουθούμε άλλη πορεία και δεν προβλέπονται κονδύλια για την ευδοκίμηση των στόχων και πώς μπορούμε αηφόρο να ακολουθήσουμε στην ΚΑΠ μακροπρόθεσμα. Τότε πρέπει κάτι να αλλάξει στο σύστημα και να έχουμε πιο αποτελεσματικές προτάσεις από ό,τι έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Ε, Μπρίτα, και μετά σε κρίσκι. Εγώ ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για το γεγονός ότι ήρθατε εδώ για να παρουσιάσετε αυτά τα θέματα. Ουσιαστικά ανταποκρίνεσαι σε αυτό το οποίο πάντα ζητούσαμε από το Ευρωκοινοβούλιο, να γίνουν περισσότερα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας για τη γεωργία. Και σε θέματα χρηματοδότησης είδαμε και προτάσεις ότι περισσότερα κονδύλια είχαμε πει πρέπει να ζητηθούν για την έρευνα και την ε, ανάπτυξη εκεί. Ερώτημα για μένα, πώς θα δημιουργηθεί η γεφυροποίηση μεταξύ αυτών των δύο τομέων, με πιλωτικά προγράμματα ή μήπως με βάση ε, εργασίας ε, που θα προσανατολίζονται στο να ανταποκριθούν σε αυτούς τους στόχους. Τι ακριβώς θα γίνει και προβλέπεται με τη στρατηγική για την διασύνδεση του Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Αλληλείας και του Ταμείου Ανάπτυξης υπαίθρου και του Περιφερειακού Ταμείου να υπάρξει διασύνδεση κομβικά Πώς θα προσεγγίσουν οι δράσεις η μία την άλλη. Εδώ πολλούς τομείς σίγουρα βλέπουμε ότι δημιουργούν επικαλύψεις και πρέπει από πλευράς χρηματοδότησης να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Ευχαριστώ. Μπρίτα και μετά Ευχαριστώ Μπρίτα μάλλον και το Σεκυριέσκη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μάθω να, μου πείτε κάτι περισσότερο για το εξή. Ε, Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα, τις πατέντες, τις νέες τεχνολογικές λύσεις ή μήπως ε, μεγαλύτερη εκβιομηχάνηση της παραγωγής. Τι θέλουμε να κάνουμε, ποια είναι η ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των μέων. Τι αντιλαμβανόμαστε με τον όρο καινοτομία, ε, κάτι που, καινοτομία που ταυτόχρονα, μια παραγωγή η οποία θα είναι ταυτόχρονα βιώσιμη περιβαλλοντικά, οικονομικά κλπ. Και τι σημαίνει καινοτομία σε αυτή τη μακρά αλυσίδα από το χωράφι έως το τραπέζι. Διότι η καινοτομία είναι διαφορετική στο χωράφι, διαφορετική στο βιομηχανία, διαφορετική στο εμπόριο. Άλλη ερώτηση. Χρηματοδότηση. Γιατί είδους χρηματοδότηση ομιλούμε στην Γεωργία υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές, ας πούμε, ε, μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις αφενός, όπου οι οποίες διαθέτουν και πόρους για έρευνα και καινοτομία και θετικά αποτελέσματα. Από την άλλη, μικρές εκμεταλλεύσεις, όπου εκεί η καινοτομία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό μικρές εκμεταλλεύσεις με φτωχούς γεωργούς οι οποίοι δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα και να υπάρξει πρόοδος σημαντική. Άρα λοιπόν τι είδους μέσα εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διαφορές. Ας πούμε καινοτομία στις μεγάλες χημικές βιομηχανίες. διότι μπαίνουν και αυτές οι μονάδες στην αγορά και διαμορφώνουν, διαμορφώνουν την εικόνα της αγοράς συνολικά. Καλώς έλεξαν οι παρεμβάσεις, οπότε θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Σιλ να δώσει κάποιες απαντήσεις που uh, Thank you for... Μάλιστα, σας ευχαριστώ για αυτές τις ερωτήσεις. Λοιπόν, υπό το σύνθημα και έννοια να ενώσουμε, συνενώσουμε τις δυνάμεις μας για να επιτύχουμε λύσεις για την βιώσιμη αηφόρο γεωργία. Πολλά μπορούν να γίνουν. Πρέπει να εφαρμόζονται όμως και να μπορέσουν να γίνουν συνολικά και όχι κατακαιρματισμένα όπως ε, μέχρι σήμερα ήδη συζητώντας μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκομένων δίνει ευκαιρία για καλύτερη στοχοθέτηση, επικέντρωση και ε, καλύτερο συντονισμό. Αυτή είναι η ιδέα μας για την ερμηνεία της ε, καινοτόμου εταιρική σχέση. Τώρα, για τι συζητήσει στα κράτη-μέλη. Ναι, πράγματι, διεξάγονται συζητήσει στα κράτη-μέλη υπό την γενική έννοια των καινοτόμων αυτών εταιρικών ε, συμπράξεων. Είχαμε πολλέ συζητήσει με ενδιαφερόμενου, εμπλεκόμενου, κυβερνητικέ αρχέ, ΜΚΟ, για την εταιρική γεωργική καινοτόμο δράση και εταιρική σχέση, η ιδέα είναι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Η αμφίδρομη δράση, οι απαντήσεις που είχαμε ήταν θετικές. Είχαν όλοι στις απαντήσεις τους τοποθετηθεί ευνοϊκά και είπαν ναι, αυτός ο στόχος αξίζει τον κόπο. Ας κάνουμε την προσπάθεια. Τώρα, γενικές εταιρικές ε, ε, καινοτόμες συμπράξεις ε, έχουν καμιά φορά κάποιες επιφυλάξεις. Το γνωρίζουμε αυτό που αντιμετωπίζουν. Στη Γεωργία έχουμε μια πιο εξειδικευμένη ξεχωριστή κατάσταση με ένα πολύ εξειδικευμένο πλήρες πακέτο μέτρων που θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία για να επιτευχθούν αποτελέσματα μέσω αυτής της εταιρικής δράσης. Αναφέρθηκα στα μέτρα συνεργασίας. Άλλα μέτρα είναι οι συμβουλές ε, προς ε, γεωργικές μονάδες εκμετάλλευσης κτλ. Πολλά μπορούν να κινητοποιηθούν με πιο στοχοθετημένο και αποτελεσματικό τρόπο. Και για τα δημοσιονομικά, τα κονδύλια, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Προπολογισμό, δημοσιονομικό πλαίσιο για τα κονδύλια που οι δράσεις που προβλέπουμε θα χρηματοδοτούνται επαρκώς. Φυσικά έχουμε τον κόσμο της υπαίθρου. Αυτό τι σημαίνει. Συνυπευθυνότητα. Οι αρχές, οι υπεύθυνε θεσπίζουν τα προγράμματά τους εξισορροπώντας ε, προτεραιότητας από κοινού με τα έγγραφα κοινή στρατηγικής δράσης. Ανταποκρινόμενοι πάντα στις ανάγκες που υπάρχουν επιτόπου. Η πείρα δείχνει ότι αν δεν ξεκινάμε επαρκώς ε, ενωρίς τις συζητήσεις ώστε να δούμε πού θα είναι το κέντρο βάρος, και πώς θα ερμηνευθούν για την επίτευξή τους οι στρατηγικοί στόχοι υπάρχει ο κίνδυνος απλά και μόνο να μετεξελίσσονται κάποια προγράμματα αντί να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες και οι προκλήσεις. Ακριβώς αυτό είναι το νόημα λοιπόν της εταιρική καινοτόμου δράσης ως εταιρική σύμπραξης. Να μπορέσουμε καινοτόμα να δράσουμε στόχοθετημένα για την επίτευξη στόχων αποτελεσματικά. Αυτό είναι αηφορία, δια, τηρώντας και διασφαλίζοντας τους φυσικούς πόρους και τις παραγωγικές δυνατότητες και διεργασίες. Είναι θέμα αηφορίας, οικονομικής και βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας. Όλοι γνωρίζουμε ότι μόνο μια γεωργία που είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική, που μπορεί να, ο γεωργός να εισπράξει αρκετά για το εισόδημά του για να επιβιώσει, μόνο μια τέτοια γεωργία μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να επιβιώσει. Έχουμε και πολιτικές και έχουμε μια ξεχωριστή κατάσταση που δημιουργείται και για την ε, γεωργία Αυτά όλα μπορεί να δημιουργούν κάποιες διαφοροποιήσεις και διαφορές όσον αφορά τις άλλες εταιρικές σχέσεις για καινοτομία στην Ευρώπη. Αν δει κανείς τις δυνατότητες για την ε, ενεργό γύρανση υπάρχουν διαφορές. Το θέμα μας είναι όχι μόνο να επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα αλλά να διευρύνουμε το πλαίσιο συζήτησης. Να ληφθούν υπόψη τα αιτήματα, οι ανάγκες, οι εξειδικευμένες ανάγκες των χρηστών για, αυτές τις, ε, ε, για αυτούς τους που έχουμε θέσει. Ίσως έτσι θα μπορέσουμε να διαφοροποιήσουμε και να μορφοποιήσουμε τις δράσεις μας πιο ενεργά και αποτελεσματικά από ότι αν μείνουμε μόνο σε επιφυλάξεις και δισταγμούς. Πώς θα υπάρξει γέφυρα μεταξύ επιστήμης και γεωργικής πρακτικής, αγρονομικής πρακτικής. Πρέπει να δούμε βέλτιστες πρακτικές να υιοθετηθούν σε σχέση με τις ε, προτάσεις ε, που έχουμε, ε, που υποβάλλονται προς εκτέλεση. Η πείρα δείχνει ότι αυτό μπορεί να είναι είναι μια πηγή αποτελεσματικής δράσης, ανταλλαγή βιωμάτων και εμπειρίας, αλλά και διατομεακά, διακλαδικά να μπορέσουν να συμπράξουν οι εμπλεκόμενοι, ώστε να υπάρξουν κίνητρα για ομάδες και ε, πρωτοβουλίες για να είμαστε αποτελεσματικοί. Υπό τον όρο ότι θα υπάρξει αυτό το ευέλικτο μέσο ε, διατομεακά, διακλαδικά, 4-5 γεωργοί και σύμβουλοι, επιστημονικοί σύμβουλοι, να μπορούν να συνέρχονται ώστε να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα ζητήματα εξειδικευμένα σε κάποια μονάδα εκμετάλλευσης, γεωργική μονάδα, έτσι, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο διασύνδεσης και διαδικτύωσης θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτή την ανταλλαγή ροής πληροφοριών και κάτι τελευταίο, η έννοια της εταιρικής καινοτόμου δράσης και σύμπραξης. Μας κάνει να πούμε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά τις διαφορές και διαφοροποιήσεις και όσον αφορά και την τεχνολογία και τις δυνατότητες χρήσης στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι περιοχές παραδοσιακής γεωργίας. Δεν είναι υποχρεωτικά η πιο καλή ιδέα να προβλέπει κανείς μία εξέλιξη επαναλαμβάνοντας ε, τα ίδια σφάλματα του παρελθόντος ε, χωρίς να υπάρξουν αλλαγές. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη, αυτό είναι διαμφισβήτο. Αλλά θα πρέπει να βρούμε τη σωστή προσέγγιση ευθύ εξ αρχής. Πώς αυτή η ανάπτυξη μπορεί να γίνει με το πιο ανταγωνιστικό, οικονομικά υγιή και πιο αηφόρο ε, ανταγωνιστικό τρόπο. Έχουμε συνειδητοποιήσει τις διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά το επίπεδο ανάπτυξης και πρέπει να προσαρμοστούμε και να αντιμετωπίσουμε εντοπίσουμε αυτές τις ανάγκες και όσον αφορά και την ανάπτυξη, την έρευνα και την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί που πρέπει να είναι πάντα καλά προσαρμοσμένη στις ανάγκες και διαφορετικές δομές. Νομίζω κάλυψα όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Σιλ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτών των δύο ημερών. Καθορισμός των εισηγητών σήμερα το πρωί Στη συνεδρία των συντονιστών πήραμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις και τις εκθέσεις που πρέπει να κάνει η Επιτροπή μας. Σας ενημερώνω ότι σήμερα το απόγευμα είναι σημαντική αυτή η συνεδρίαση της Πολωνικής Προεδρίας. Θα είναι εκεί επίτροπος παρούσα. θα συμμετάσχουν πολλοί από εσά στη, συζήτηση και στο τέλος σας δίνω ραντεβού για τις 19 Δεκεμβρίου στις 3 το μεσημέρι, 3 το απόγευμα και στις 20 Δεκεμβρίου από 9 το πρωί μέχρι τις 12.30. Αυτές είναι οι επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ όλους και είστε επανειδήν. Θα λέμε το απόγευμα. Γεια σας.